Colleagues, can I Ας αρχίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι και την απογευματινή μας συνεδρίαση με ιδιαίτερη χαρά. Σας παρουσιάζω τον Υπουργό Συγκεβίσιους. Ελπίζω να προφέρω καλά το όνομά του. Είναι Λιθανός Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Προεδρεύων του Συμβουλίου ο οποίος και θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας. Συνεπώς, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία μαζί σας και με την Προεδρία σας για το επόμενο εξάμεινο. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Πρόεδρε, είναι ιδιαίτερη χαρά και προνόμιο για μένα να μπορώ να δεχτώ την πρόσκλησή σας και να έρθω να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας. Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα της χώρας μας τα τελευταία 23 χρόνια, από τότε δηλαδή που κερδίσαμε την ανεξαρτησία μας. Νιώθουμε συγχρόνω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη τώρα που αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου. Είμαστε όμως πεπισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε. Ότι θα μπορέσουμε δηλαδή αποτελεσματικά και αποδοτικά να φέρουμε σε πέρα στο έργο μας. Τους επόμενους έξι μήνες θα επικεντρωθούμε σε επικοδομητικές συνομιλίες με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εξεύρουμε πρακτικές λύσεις και να έχουμε έτσι απτά αποτελέσματα υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνετε ευκαιρία τώρα στην αρχή της Προεδρίας μας να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητές μας και να συζητήσω μαζί σας διάφορα σημαντικά ζητήματα. Η Επιτροπή σας θα ασχοληθεί με πολλά σημαντικά θέματα το επόμενο εξάμεινο. Πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή λοιπόν είναι μια ευκαιρία για να θέσουμε τα θεμέλια για καλή συνεργασία ανάμεσα στην Προεδρία μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού. Η εμπιστοσύνη και η συνεργασία είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα, παρά δηλαδή την οικονομική κρίση και τις διάφορες προκλήσεις που τη συνοδεύουν. Η λιθωνία λοιπόν θα επικεντρωθεί σε μέτρα τα οποία θα προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και θα διασφαλίσουν και δημοσιονομική σταθερότητα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι τώρα που πλησιάζουμε και στις επόμενες ευρωεκλογέ που προβλέπονται για το Μάιο του 2014, είμαστε πιο κοντά και στην ε, λήξη της ε, θητείας σας και του νομοθετικού σας συνεπώς έργου. Γι' αυτό και θέλετε να προχωρήσετε όσο γίνεται περισσότερο και να καταλήξετε ή όσο γίνεται περισσότερες νομοθετικές προτάσεις, κάτι το οποίο περιμένουν βέβαια και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέα προνόμια και αρμοδιότητες και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα κατάσταση. Και γι' αυτό όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που διαπιστώνουν τη νέα πραγματικότητα πρέπει συγχρόνως να διασφαλίσουν ότι οι δράσεις τους και οι αποφάσεις τους φροντίζουν για να προχωρήσει με ήπιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μην ξεχνάμε ότι οι πολίτες μας παρατηρούν και περιμένουν από μας αποτελέσματα. Άρα λοιπόν πρέπει να τους προσφέρουμε αποτελέσματα. Και πάνω απ' όλα η Λιθουανία κατά τη διάρκεια της προεδρίας της θα προσπαθήσει να πετύχει πράγματι αποτελέσματα και ξέρω ότι ο κόσμος θα μας κρίνει ανάλογα με το πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρωτής της σημασίας. Οι συνάδελφοι και εγώ, προετοιμάζοντας την ε, Προεδρία, καταλήξαμε ότι είναι προτεραιότητά μας οι καλές μας σχέσεις μαζί σας. Γιατί ό,τι οι ανταλλαγές απόψεων είχαμε μέχρι τώρα μαζί σας ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικές. Θέλουμε λοιπόν έτσι να βρεθούμε πιο κοντά στο Κοινοβούλιο και να προετοιμαστούμε έτσι από την πρώτη μέρα της Προεδρίας μας για το έργο μας. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή θα βαθύνει ακόμα περισσότερο τους υπόλοιπους μήνες της χρονιάς αυτής. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους προκατόχους μας, τους Ιρλανδούς δηλαδή, την Ιρλανδική Προεδρία. Ο κύριος Λίο Βατκάρ και οι συνεργάτες του αποδείχθηκαν εξαίρετοι συνάδελφοι. Πρόκειται για μια Προεδρία η οποία κατάφερε πολύ σημαντικά επιτεύγματα και σίγουρα έβαλαν τον πύχη πολύ ψηλά για μας. Ό,τι αμφιβολίες μπορεί να είχαμε για τις προτεραιότητες όσον αφορά τις μεταφορές, δεν υπάρχουν πια μετά από τη συνάντηση που είχα μαζί σας κύριε Πρόεδρε, γιατί εσείς και οι συνάδελφοί σας στην Επιτροπή αυτή εκπροσωπείτε έναν τεράστιο, είσαστε μάλλον αποτελείτε ένα τεράστιο πλούτο γνώσης και εμπειρίας σε θέματα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν για μας είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε από τις δικές σας ιδέες και ανησυχίες. Αυτή, αυτού του είδους λοιπόν ειλικρινείς ανταλλαγές απόψεων θα συνεχιστούν, να ξέρετε, με θετικό πνεύμα και στο μέλλον. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων της Ιρλανδικής Προεδρίας, του κυρίου Λέο Βάρατκαρ δηλαδή, που ήρθε μάλιστα και στην Επιτροπή σας τον προηγούμενο μήνα, ήταν ο κανονισμός για τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ο κανονισμός για την διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, Connecting Europe. Πρόεδρε, μαζί με τον κύριο Βαρατκάρ και εσάς, πιστεύω ότι κάνουμε σημαντική δουλειά. Μετά το αποτελέσμα της Ιρλανδικής Προεδρίας, η πρόταση αυτή θα προχωρήσει και θα έχει αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Επειδή θέλουμε μια ανοιχτή Ευρώπη επίσης, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε δίκτυα υποδομών φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών, την οδική ασφάλεια και την διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικτύων μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε μια γενική προσέγγιση όσον αφορά την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο και να δημιουργήσουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον, να αυξήσουμε επίσης και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα προσπαθήσουμε συγχρόνως να συμφωνήσουμε για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον κανονισμό για την ε, υπηρεσία της ευρωπαϊκής δορυφορικής πλοήγησης κάτι που πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Τώρα, το τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό γιατί σε πήγες μεταφορές. Στόχος είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων και έτσι μπορούμε να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε τα τεχνικά θέματα που αφορούν το πακέτο αυτό και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια γενική προσέγγιση για, το, για την οδηγία όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Θέλουμε επίσης να προδεύσουμε και σε σχέση με τον κανονισμό για, την, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Θα έχουμε μάλιστα ένα σεμινάριο με επιχειρήσεις ε, από τους Ευρωπαϊκούς Σιδηροδρόμους σήμερα το βράδυ και εκεί θα δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές ε, διασυνοριακές μεταφορές. Και ο κύριος Ζήλη συμφώνησε να έρθει και ελπίζω να έρθουν και άλλοι από εσά σήμερα το βράδυ. Έρχομαι τώρα στο πακέτο το σχετικό με την αξιολόγηση των ε, οδών, των οδικών αρτηριών. Οι προπτικές της συνεργασίας και επίτευξης συμφωνής για το πακέτο αυτό είναι σημαντικές. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία με τους εισηγητές σας και την κυρία Σενάλοβα και τον κύριο Κούν και την κυρία Σάφη Αρτούμαστ. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του επί των τριών προτάσεων του πακέτου αυτού και την προηγούμενη εβδομάδα το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δικιά του θέση. Συμφωνία για προτάσεις όσον αφορά περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων, ελέγχους ε, στους δρόμους των εμπορικών οχημάτων και τα έγγραφα κα... καταχώρησης οχημάτων είναι και αυτά ένα σημαντικό βήμα προς την οδική ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα την αεροπλοεία. Υπάρχει πρόοδος στο Συμβούλιο προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιριών και έχουμε συζητήσει και τα θέματα των αποζημιώσεων σε περίπτωση ακυρώσεων, καθυστερήσεων ε, ή άρνησης επιβίβασης σε κάποιον επιβάτη. Ελπίζουμε να πετύχουμε μια κοινή προσέγγιση τελικά τον Δεκέμβριο. Και ευχαρίστω να αρχίσουμε συζητήσεις για τα θέματα αυτά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόλο που οι κύριες συζητήσεις για αυτό το θέμα θα γίνουν σίγουρα επί ελληνικής προεδρίας. Θέλουμε επίσης να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσει μαζί σας σχετικά με τον κανονισμό όσον αφορά την αναφορά συμβάντων στην πολιτική αεροπορία. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με την εισηγήτρια, την κυρία Βεϊράκ. Ξέρουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η πρόταση αυτή. Διότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών. Επίσης, να ξέρετε ότι θα ζητήσω από τους αδέρφους μου υπουργού να εγκρίνουν στο Συμβούλιο την απόφαση για το ΣΕΖΑΡ. Το Συμβούλιο θα αρχίσει επίσης να συζητάει το θέμα του ενιαίου ουρανού 2. Στις 16 Σεπτεμβρίου, στο Βίλνιους μάλιστα, να ξέρετε ότι έχουμε μια άτυπη συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών, όπου θα προτείνω να συζητήσουμε την πρωτοβουλία αυτή για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Ο κύριος Κάλλας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποσχέθηκε ότι θα έρθει. Και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να δω εκεί και τους εισηγητές και από την Οικονομική ε, Επιτροπή, την κύριο Γιάτ Ελπίζω και εσείς κύριε Πρόεδρε και άλλα μέλη της Επιτροπής σας να έρθετε επίσης. Στον τομέα τώρα των θαλασσίων μεταφορών. Εδώ θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια προσέγγιση του Γενικού Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για την πολιτική χρηματοδότηση του, οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Πρόκειται για οργανισμό που συζητάει τα θέματα της ρήπανσης μεταξύ άλλων από πλατφόρμες ε, πετρελαίου. Θέλουμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Με τη βοήθεια του κύριου Τέιλορ θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ώστε απρόσκοπτα να μπορεί να λειτουργήσει ο οργανισμός και η συμφωνία αυτή προβλέπεται για το 2014. Θέλουμε επίσης να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις μαζί σας και για τον θαλάσσιο εξοπλισμό, τη σχετική οδηγία δηλαδή, προκειμένου να διασφαλίσουμε μια πρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα του θαλάσσιου εξοπλισμού. Θέλουμε επίσης υψηλό επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα και αποφυγή ρήπανσης. Προσβλέπουμε σε επικοδομητική συνεργασία μαζί με τον εισηγητή σας και αντιπρόεδρο, τον κύριο Ρίκε. Επίσης, θέλουμε να προχωρήσουμε και σχετικά με το πλαίσιο πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών λιμένων και διαφάνεια επίσης όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές των λιμένων τον Οκτώβριο η Λιθουανία, στη Λιθουανία μάλλον θα γίνει μια συνάντηση σε 9 Οκτωβρίου των Υπουργών από την Ανατολική Εταιρική Σχέση Υπουργών Μεταφορών. Είναι πολύ καλό γιατί θα συζητήσουμε και με τρίτες χώρες για θέματα υποδομών μεταφορών. Θα μπορέσουμε έτσι να συζητήσουμε για την διασύνδεση των ευρωπαϊκών δικτύων με Κίνα των έξι χωρών που γειτονεύουν με μας. Πιστεύω ότι σχετικά προγράμματα έχουν τεράστια αξία. Τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής θα παρουσιαστούν στην διάσκεψη που θα έχουμε στο Βίλνιους επίσης τον Οκτώβριο. Τώρα επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητές μας στον τομέα του τουρισμού. Παρόλο που πρέπει να παραδεχτώ εδώ ότι την ευθύνη για τον τουρισμό στην Λιθουανία τον έχει ο συνάδελφός μου υπουργό Οικονομικών. Παρ' όλα αυτά ευχαρίστω να μιλήσω εδώ και εκ μέρους του. Ο τουρισμός ασφαλώς και αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, οικονομικής δραστηριότητας γιατί ενισχύει την απασχόληση και το επιχειρίζεστε. Εφόσον υπάρχει ανάπτυξη στον τουρισμό, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για ολόκληρη την Ευρώπη. Η Λιθουανία το ξέρει αυτό. Οπότε θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ευκαιρίες για τον τουρισμό προκειμένου να ενισχυθεί ο τουρισμό στην Ευρώπη. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Λιθουανία λοιπόν οργανώνει το 12ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον τουρισμό στο Βίλιο, 17 και 18 Οκτωβρίου. Ο τίτλος θα είναι «Τουρισμός ω παράγοντα οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική αλλαγή και ευημερία. Το φόρουμ αυτό λοιπόν θα εξετάσει δυνατότητες συνεργασίας, ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού. Θα συζητήσουμε επίσης για τη φορολόγηση των ε, τουριστικών επιχειρήσεων. θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τον Παγκόσμιο Τουρισμό θα έχουμε και τουριστικές ε, ενώσεις από την θάλασσα της Βαλτικής. Ελπίζουμε ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε χρήσιμες ιδέες και θα διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη θα εξακολουθεί να είναι η πιο ελκυστική περιοχή για τον τουρισμό. Κύριε Σίμψον, χαιρόμαστε πάρα πολύ που δηλώσατε ότι θα συμμετάσχετε στο φόρουμ αυτό. Ευχαρίστω να σας υποδεχτούμε στη χώρα μας. Το επόμενο εξάμεινο θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη σχέση μας με εσάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι μπορούμε αποτελεσματικά να πετύχουμε την ισορροπία και καλές λύσεις. Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος εξαρτάται από τον άτυπο διάλογο που γίνεται ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και εφόσον τηρούνται οι κανόνες που υπάρχουν και έχουν αποδεχθεί τα δύο αυτά όργανα. Κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας λοιπόν θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την παράδοση συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. Προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ό,τι ερωτήσεις έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Εκτός από τους ε, συντονιστές εδώ τον κύριο Μπακ, Σάβησαν και Κούν. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Κούτζιας, Κόλλη, Τάνζα. Να ρωτήσω καλύτερα ποιος δεν θέλει να μιλήσει. Οι συντονιστές πρώτα και εσείς πέφτετε σε αυτήν την κατηγορία κύριε Κόλτσεκ. Είπαμε Φιντάντσα, Μπένιον, εντάξει. Τρία λεπτά για τους συντονιστές και δύο λεπτά για τα μέλη. Κύριε Γκρός, έχετε τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Συγγνώμη που ήρθα ε, κάπως καθυστερημένα και δεν πρόλαβα να ακούσω όλα αυτά που είπατε. Θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι έρχεστε από μια σημαντική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Βαλτική και ελπίζω να είναι πραγματικά σημαντική προεδρία σας. Τρία κεφάλαια σημαντικά. Το ένα είναι η εφαρμογή των μέτρων αυτό είναι κάτι που δεν το αναφέρει πάντα το Συμβούλιο, γιατί για πολλοί τομεί καθυστερούν τα πράγματα και έχουμε σαν παράδειγμα ότι η Κομισιόν χρειάστηκε να αλλάξει τη διατύπωση της πρότασης για τους ενιαίους εθέρες, γιατί η προηγούμενη διατύπωση δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί σε επίπεδο που περιμέναμε. Θα χαιρόμαστε λοιπόν ε, αν δίνατε μια προτεραιότητα στο θέμα αυτό και με την ε, επισήμανση τουλάχιστον από την ε, πλευρά μας δεν μπορεί ότι δεν μπορεί το Συμβούλιο να αποφασίσει μαζί με τα κράτη-μέλη και μετά να δει ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά που έχουν αποφασιστεί. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Όταν μιλάμε για το τέταρτο πακέτο για τα σιδηροδρομικά και εδώ υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία χρονίζουν και υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες σε σχέση με το θέμα αυτό. Θα χαιρόμαστε λοιπόν να προωθηθούν συζητήσει για τη διαλειτουργικότητα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο και ως Συμβούλιο ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο επιμένει να μείνουν όλα αυτά τα θέματα στα επίπεδο μιας δέσμης. Λοιπόν, η αποτελεσματικότητα θα επιτευχθεί αν τηρηθούν όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση και όχι αν ακολουθηθεί ο δρόμος της μικρότερης αντίστασης. Στον τομέα των οδικών συμπεριφορών θέλουμε να λάβετε το περιεχόμενο υπόψη των τριών εκθέσεων για την ασφάλεια, η επιτόπιοι έλεγχη και τα άλλα θέματα. Επίσης είναι σημαντικά τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτά δεν είναι θέματα τόσο τεχνικά όσο τα άλλα. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια πρόοδος. Κάτι ακόμα, μια α, ε, αίτηση προς εσάς και δεν είμαστε ίσως η μόνη ομάδα που ζητάει κάτι τέτοιο. Μετά από πολλές και δύσκολες συζητήσεις καταφέραμε να κλείσουμε τις τρεις εκθέσεις για τα θέματα του εναέριου χώρου και των υπηρεσιών και να έχουμε μια γενική στάση στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για την ηχορύπανση, για τα σλότς, τις χρονοθυρίδες και την εξυπηρέτηση εδάφους. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει μια πραγματική προσπάθεια να μην περικλέψει τα πράγματα. Κάντε μας λοιπόν τη χάρη να δεχτείτε τα θέματα αυτά να παραμείνουν από κοινού σαν πακέτο, γιατί και εμείς χρειάστηκε να ξεπεράσουμε πάρα πολλές αντιδράσεις και έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια για να παραμείνει το πακέτο αυτό πακέτο μια δέσμη μέτρων. Σας ευχόμαστε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και βασιζόμαστε σε εσάς. Κύριος Καδράουι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή σας. Και εγώ σας εύχομαι εκ μέρους της ομάδας μου κάθε επιτυχία το επόμενο εξάμεινο. Είναι πράγματι η πρώτη προεδρία της χώρας σας. Και μπορώ να σας πω ότι έχετε μεγάλη ευθύνη στους ώμους σας, αλλά να ξέρετε ότι ίσως είναι η τελευταία προεδρία η οποία θα μπορέσει να ολοκληρώσει κάποιες νομοθετικές υποθέσεις. Φυσικά μετά ακολουθεί και η ελληνική προεδρία, αλλά θα έχουμε τότε τις ευρωεκλογέ, οπότε Μάρτιο, Απρίλιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε πολλές δυνατότητες να προωθήσουμε την νομοθετική διαδικασία. Άκουσα το πρόγραμμά σας, περιλαμβάνει πολλά σημαντικά ζητήματα και χαίρομαι που ήδη σήμερα είχαμε την πρώτη, τον πρώτο διάλογο μεταξύ μας για τα διάφορα πακέτα και για την ασφάλεια κλπ. Είναι πολύ σημαντικό που τόσο γρήγορα αρχίζουμε. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία μέσα στους επόμενους μήνες. Ίσως να μην είναι όμως τόσο καλό. Είναι οι υποθέσεις που έχουμε σχετικά με την αεροπορία. Εδώ υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες με το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι εδώ και χρόνια έχουμε γκρίνει κάποια νομοθεσία και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε πιο αποτελεσματικά μέτρα. Ξέρετε όμως ότι στην πράξη δεν έχουν γίνει πολλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε με νέα πρόταση. Γι' αυτό και θέλω να κάνω έκκληση να προχωρήσουμε παρακαλώ με τα πλεονεκτήματα, αυτά πλεονεκτήματα και για το περιβάλλον και για τους καταναλωτές, για όλους μας. Το πακέτο για την αεροπορία, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι πάνω-πάνω στις προτεραιότητες και εσείς είσαστε έτοιμοι, το Συμβούλιο και εμείς είμαστε έτοιμοι, οπότε ας προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα συμφωνώ και με τον κύριο Γρός. Σημειώνουμε το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποια βήματα στα τεχνικά ζητήματα κυρίως. Εμείς βέβαια έχουμε μια διαφορετική μέθοδο. Θέλουμε να εξετάσουμε όλο το πακέτο μαζί για να μπορούμε μαζί να μιλήσουμε και να το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Τέλος για τον τουρισμό Όντω είναι ένα κλάδος που δεν πρέπει να υποτιμάται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην τον ξεχάσουμε τον τουρισμό τους επόμενους μήνες γιατί είναι σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους, η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του και την παρουσίαση του προγραμματός του, το οποίο είναι πράγματι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνετε την Προεδρία, μια μεγάλη πρόκληση βέβαια και ιδίως γιατί την αναλαμβάνετε στο τέλος μιας νομοθετικής περίοδου που είναι πολλά τα θέματα, τα νομοθετικά τα οποία θα πρέπει να περατωθούν. Φυσικά και η Ιρλανδική Προεδρία έχει βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά έχετε αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικά πακέτα μέτρων τα οποία είναι στην, ε, στα χέρια σας. Έχουμε τα εναλλακτικά καύσιμα, έχουμε το Connecting Europe, έχουμε τα δίκτυα των υποδομών τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όλα αυτά έχετε τονίσει και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι επειδή έρχομαι από την ε, Γερμανία που βρέχεται εν μέρη από τη Βαλτική με, ενδιαφέρεται, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η δημιουργία της υποδομής στην Βαλτική. Μίλησατε και για το σιδηροδρομικό πακέτο εμείς το συζητήσαμε αυτό, υπάρχουν πολλά προβλήματα και το πακέτο για τα θέματα οδικής ασφάλειας έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και είναι έτοιμο για απόφαση. Σε ό,τι αφορά την ε, αεροπορία, μιλήσατε για τα δικαιώματα των ε, πολιτών και τα συμβάντα στον εναέριο χώρο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολα. Για μας είναι σαφές ότι δεν είναι καθόλου εύκολα, αλλά και πάλι σας λέω ότι δεν μπορείτε εσείς να αποφασίσετε, θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα αυτά να προχωρήσουν. Δεν μπορεί να έχουμε μια ε, εναρμόνιση προς τα κάτω και να μειώσουμε τις παροχές και το επίπεδο ποιότητας. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια κοινή λύση. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η αντιμετώπιση των θεμάτων του νεαρίου χώρου, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, θάλασσα και τους λιμένες, η ΕΜΣΑ λειτουργεί πολύ καλά. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το έργο της. Έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία σε σχέση με τον ναυτικό εξοπλισμό και έχουμε τώρα και τις υπηρεσίες λιμένων οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και εδώ θέλω να θέσω το, το ερώτημα αυτό. Είμαι εισηγήτρια για την ε, χωροταξία του θαλάσσιου χώρου και τα θέματα αυτά των παρακτήων περιοχών, μας ενδιαφέρει και εδώ να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και από την πλευρά του Κοινοβουλίου να λάβετε υπόψη δική μας γνωμοδότηση. Έχετε πει ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη. Αυτή η μπλε ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και γι' αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε στην χωροταξία στον χώρο αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουν να προωθηθούν όλα αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της Λιδανικής Προέδρειας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ, τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, Σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σα και εγώ φυσικά θα σα ευχηθώ κάθε επιτυχία εξ ονόματο των Πρασίνων τη ομάδα μου για την περαιτέρω εργασία σα. και θέλω να σα καλωσορίσω όχι μόνο εσά, αλλά και τη χώρα σα η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το έλεγε κάποιος αυτό πριν από 25 χρόνια θα το λέγανε θεότρελο, αλλά σήμερα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ελέγχθησαν πάρα πολλά, εγώ θα ήθελα να τονίσω μονάχα δύο σημεία. Η ενία η ευρωπαϊκή εθέρες. Δεν είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Έχουν κλείσει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια πραγματικότητα. Από την 1η Οκτωβρίου του 2012 θα πρέπει να ισχύουν όλα αυτά. Το ξέρανε τα κράτη-μέλη. Παρόλα αυτά αντιστέχονται και παραβιάζουν την ομοθεσία που έχουν εγκρίνει τα ίδια κράτη-μέλη. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση win-win. Μπορούμε να μειώσουμε τον προσωπικό στον ενάριο χώρο, να έχουμε λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Επομένως όλα αυτά μπορεί να είναι θετικά και τα μπλοκάρει το Συμβούλιο. Σας παρακαλώ λοιπόν το Συμβούλιο να κάνει τα απαραίτητα για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει κράτος δικαίου στην Ευρώπη και ο νόμος εφαρμόζεται. Δεύτερον, εγώ έχω εκλεγεί το 2004 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 2003 ήρθα από, πήγα από το Βερολίνο όπου ήμουνα στην Ταλίν. Εννιά φορές άλλαξα τρένο στα σύνορα Λετωνίας-Εστονίας πήγα με τα πόδια από τον ένα σταθμό στον άλλο. Μετά από πολλές ώρες είδα ότι υπήρχαν και ατμομηχανές προπολεμικές οι οποίες με φέρανε στον προορισμό μου και το όλο ταξίδι κρότησε 27 χρόνια. Αν μπορέσετε λοιπόν να περάσετε το συνδρομικό πακέτο, αυτό θα είναι μια μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. Μόλις εξελέγην, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να μπορέσουν τα θέματα αυτά της Βία Μπάλτικα μέσα στα πιο σημαντικά θέματα προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία προχώρησαν αλλά όχι ε, επαρκώς. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα σε εσά. Εφόσον δεν γίνεται τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κάνετε μια περαιτέρω προσπάθεια. Θα πρέπει να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις, θα πρέπει να πείσετε τα τρία βαλτικά κράτη και την Πολωνία να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Εμείς δεν θέλουμε τα τρία βαλτικά κράτη να αποκοπούν, να είναι αποκομμένα από την Ευρώπη, όπως ισχύει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει νόημα να μην μπορεί να υπάρχει κυκλοφορία επιβατών μεταξύ Λετωνίας και Λιθουανίας. Θα ήθελα λοιπόν από τη δική σας πλευρά να υπάρχει μια αποφασιστική στάση και εσείς ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, συγγνώμη, αλλά και ω Υπουργό Λιθουανία να αναλάβετε και να κάνετε τι απαραίτητε ενέργειε για να πραγματοποιηθεί η Βία Ο κύριο Ζήλε για του συντηρικού και μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στην Προεδρία, διότι η Λιθουανική Προεδρία αφορά όλε τι ε, χώρε τη Βαλτική. Ε, δύο ζητήματα. Το για ε, το πακέτο στο οποίο αναφερθήκατε αναφορικά με την ε, ασφάλεια των σιδηροδρόμων και την οδική ασφάλεια αλλά και το νέα την ευρωπαϊκή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Θα ακολουθήσετε το παράδειγμα που έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση των αεροπορικών ε, μεταφορών για την ασφάλεια ή όχι. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην Βαλτική και θα είμαι ειλικρινής ε, κύριε Υπουργέ. Εμείς εδώ στο σώμα ανέκαθεν υποστηρίζαμε την ε, βελτίωση των μεταφορών των ειδικά στις χώρες της Βαλτικής, θα πρέπει να ε, προωθηθεί ως πρώτη στην προτεραιότητα. Εάν υπάρχει μεροδότηση της ε, τάξης του 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής, στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των τριών κρατών της Βαλτικής για την δημιουργία μιας ε, κοινή ε, επιχείρηση για την πρόθεση αυτού του σχεδίου. Υπάρχουν κάποιες ε, ομάδες συμφερόντων στον τομέα των σειροδρομικών μεταφορών και αυτές οι ομάδες λειτουργούν αποτελεσματικά στην πρώτη φάση της όλη διαδικασίας. Στη μεταγενέστερη φάση χρειάζεται να δημιουργούν διαφορετικοί θεσμοί για να αναλάβουν αυτό το έργο. Υπάρχει συνεργασία με τους ε, ρωσικούς υδροδρόμους και ε, γι' αυτό στις χώρες δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για, την, για το μέγεθος ε, των, της απόστασης ανάμεσα στις σιδηροτροχές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας νέος κοινός όμιλος επιχειρήσεων που θα ενδιαφερθεί σε μια τέτοια, μια τέτοια προσπάθεια. Θα μπορούσα λοιπόν κατά την Προεδρία να το προωθήσετε. Ευχαριστώ. Κύριο Κόλιτζακ, τρία λεπτά. Μεγάλη ευχαρίστηση που βρίσκομαι στο, συμπεριλαμβάνω μάλλον στον καταλόγα σας. Πάντα συμπεριλαμβάνεστε παρατηρία πρόεδρο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τσεχικά, παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Κύριε Υπουργέ, έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Μιλήσατε για τον τουρισμό και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για τη χώρα σας, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει από τουριστικής σκοπιάς, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω ότι πιστεύετε για τις εσωτερικές μεταφορές και την ανάπτυξή τους. Το, το, ανάπτυξη του τουρισμού για μένα είναι πολύ σημαντικό θέμα για κάποιες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως αυτό να είναι και μια προσδοκία για τη χώρα σας. Και ένα δεύτερο ερώτημα αφορά τις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Ε, πιθανότητες ε, βλέπετε να υπάρξει πόρος σημαντική διότι υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τις μεταφορές και ένα από αυτά είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση. Τώρα για τις αεροπορικές μεταφορές υπάρχει μια δέσμη, ένα πακέτο αλλά σε ό,τι αφορά τώρα τις, ε, τις, ε, τις παροχές υπηρεσιών ε, όπως και τα σλότ αλλά και τον θόρυβο που προκαλούν τα αεροσκάφη δεν μπορούν να επιληθούν φυσικά όλα αυτά δια Τώρα για τις οδικές μεταφορές συνεχίζουμε να μιλάμε για τους διαδρόμους, για τις υποδομές, για την διευκόλυνση Connecting Europe. Πιστεύετε ότι σε αυτόν τον τομέα που είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένος, ειδικά σε ό,τι φορά τα οδικά ατυχήματα, μπορείτε να προτείνετε κάποιες λύσεις όπως το θέμα του κοινού αριθμού βοήθειας 112 και για σύνδερο δρόμους και το τέταρτο πακέτο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς θα το εξετάσετε. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στα υπόλοιπα μέλη. Ο κύριος Μπακ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Πρόεδρε του Συμβουλίου. Και εγώ φυσικά θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της Λιτουανικής Προεδρίας και για το φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο μας έχετε παρουσιάσει και τους στόχους σας. Έχετε μιλήσει για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο και το χαιρετίζω ιδιαίτερα. Θα ήθελα να περιοριστώ σε δύο ή τρία σημεία. Αναφέρθηκε ήδη το θέμα του σιδηροδρομικού πακέτου θέλω να σας ρωτήσω εδώ αν θα προσπαθήσετε και πάλι να το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα ως πακέτο ή αν θα ακολουθήσετε το δρόμο του παρελθόντος και να επεξεργαστείτε μόνο τα τεχνικά θέματα. Εγώ είμαι συγητής για τα κοινωνικά θέματα που έχουν να κάνουν το πακέτο στην Κοινωνική Επιτροπή και νομίζω ότι πρέπει να διαμορφώσουμε μια κοινή άποψη και για μένα οι κοινωνικές ε, συνθήκες θα πρέπει να συνδεθούν με τον κανονισμό περί υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, PSO. Ως επίσης και εισηγητής για τα δικαιώματα των επιβατών, χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι έχετε αποδώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό και θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Βέβαια, είχα ήδη συζητήσει για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο έχετε μια γενική κατεύθυνση που θα ακολουθήσετε για τα θέματα αυτά. Ποιο είναι το πνεύμα με το οποίο εσείς θα αντιμετωπίσετε αυτό το νομοθέτημα. Και μετά μιλήσατε και για τα θέματα διαλειτουργικότητας μεταξύ των ε, διαφόρων φορέων μεταφοράς ένθεν και εκεί δεν των συνόρων. Θα ήθελα όμως να μου πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο για τα θέματα αυτά, αν είναι δυνατό, γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο μέλλον. Θα είναι σημαντικό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαβισά για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή και καλή τύχη στους γειτονές μας εύχομαι. Πιστεύω πράγματι ότι οι βαλτικές χώρες μεταξύ τους είναι σαν αδερφές. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συντονιστές, οπότε μπαίνω στην ουσία. Παρακολούθησα προσεκτικά την εισαγωγή σας. Θα ήθελα να ακούσω, μάλλον χάρηκα που άκουσα τα λόγια που είπατε από την καρδιά, όπως τα νιώθουμε και εμείς. Δεν άκουσα όμως τίποτα για το Rail Baltica, που αφορά τις βαλτικές χώρες. έχει να κάνει με τον ε, διάδρομο μεταφορών σε ένα κομμάτι της Ευρώπης, αν μη τι άλλο. Πριν από τρεις μήνες, οι τρεις πρωθυπουργοί αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτήν την κοινοπραξία κατά κάποιο τρόπο. Και να ενστερνιστούν έτσι το σχέδιο αυτό για τον διάδρομο της Βαλτικής. Όμως η λιθουανική κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται και εσείς ο ίδιος φρενάρατε το όλο σχέδιο λόγω δυσκολιών χρηματοδότησης στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί όμως, τι μπορούμε να κάνουμε για να ελευθερώσουμε το πρόγραμμα και να προχωρήσει. Ευχαριστώ κυρία Συναλόβα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε αξιότιμε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Όπως έχουμε ήδη πει εδώ, είμαι και εγώ εισηγητής ενός κομματιού του πακέτου που έχει να κάνει με, τις τεχνικές, με τους τεχνικούς ελέγχους. Ξέρω ότι σήμερα υπήρξε ήδη μια άτυπη συνάντηση με τους άλλους εισηγητές, οπότε σας ευχαριστώ που αναλαμβάνετε δράση εκ μέρους της Λιθουανικής Προεδρίας και προσβλέπω και εγώ σε στενή συνεργασία μεταξύ μας. Ελπίζω να καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμφωνία μέσα στο εξάμεινο αυτό. Πάντως πρώτα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ασφάλεια στις μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας και την ιδέα των ενιών μεταφορών, κάτι στο οποίο θα καταλήξουμε με την νομοθεσία αυτή. Έχω όμως κάποια ερώτηση για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο εγκρίναμε ένα ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική μας για να μειώσουμε τα σοβαρά ατυχήματα στους δρόμους της Ευρώπης. Κάτι που θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτό είναι και το σύστημα του ευρωπαϊκού νούμερου για κατεπήγοντα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κούν. Συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ. Σας ε, συγχαίρω και σας ε, καλωσορίζω στην πρώτη σας Προεδρία. Πιστεύω ότι και τα μικρά κράτη-μέλη έχουν παίξει ένα ιδιαίτερο ρόλο για να επιτευχθεί συμφωνία σε σημαντικά θέματα όπως ε, για το αεροπορικό πακέτο και μπορούν επομένως να προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως αυτά που είπατε ε, ανέφεραν και το θέμα των περιοδικών ε, οδικών ελέγχων και επίσης την τον έλεγχο κταίω των αυτοκινήτων. Η Λιθουανία δεν είναι μια σιδηροδρομική δύναμη, είναι μια χώρα περισσότερο θαλασσοπόρων και θέλω να σας καλωσορίσω για αυτά που θέσατε για την ναυτική ασφάλεια, για τον καλύτερο εξοπλισμό των πλοίων, για την τυποποίηση του ναυτικού εξοπλισμού σε ό,τι αφορά τα μέσα διάσωσης και ασφαλείας και την εφαρμογή των συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Επίσης όμως και τα συστήματα πλοήγησης με δορυφόρο, ε, όπως είναι ο Γαλιλαίος που είναι έτοιμα για εφαρμογή και αυτά είναι θέματα, αυτά είναι μέσα τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ασφάλεια στη θάλασσα. Άμα δει κανεί την Βαλτική που είναι μια εσωτερική θάλασσα με μεγάλη κυκλοφορία πλοίων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιωθεί εκεί η ασφάλεια με τις ε, ε, με τη δορυφορική πλοήγηση, η Λιθουανία με την Κλαϊπέδα και την σύνδεση με την Πολωνία. Όλα αυτά τα μέρη νομίζω ότι είναι χώροι που έχουν αναπτύξει και στο παρελθόν πολύ καλή συνεργασία και ελπίζουμε ότι θα τη συνεχίσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κούγκια για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς όρισατε κύριε Υπουργέ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Πραγματικά δεν σας ζηλεύω, ειλικρινά. Διότι στην θέση σας οποιοδήποτε θα είχε τα χέρια που θα του έτρεμαν. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, λίγος ο χρόνος, διάθεσή σας και πολλοί φάκελοι που έχουν τύχει επεξεργασίας και απαιτούν να προωθηθούν και να ολοκληρωθεί για να μην μην αρχίσετε να τρέμετε περισσότερο, δεν θα προσθέσω κάποιου άλλου φακέλου, κάποια άλλα ζητήματα. Θέλω να υπενθυμίσω μερικά από τα θέματα που έδειξαν οι συνάδελφοι. Καταρχήν το δέσμι για τα αεροδρόμια. Εμείς εργαστήκαμε πάνω στο ζήτημα και στην Ολομέλεια καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Εάν αληθεύει το ότι η Προεδρία θα πρέπει να εξετάζει κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να προωθεί και να ολοκληρώνει, αλλά ταυτόχρονα έχει την υποχρέωση να δώσει μια συνέχεια στις εργασίες που έχουν ήδη γίνει και εδώ βρισκόμαστε σε καταληκτική φάση. Λοιπόν, η ερώτησή μου έχει ως εξής. Προτίθεστε εσείς, αν όχι να ολοκληρώσετε, αλλά να βάλετε στη τροχιά το ζήτημα που αφορά τα αεροδρόμια. Δεύτερο, ο τουρισμός. Για χρόνια λέγαμε ότι ο τουρισμός είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη και για να δώσουμε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτή την παραπάνω ταχύτητα για να εξέλθουν από αυτήν την ε, οικονομική κατάσταση που επηρεάζει τις χώρες μας. Το δεύτερο δεν αποτελεί ερώτηση. Πριν αρχίσει να χτυπάει το σφυράκι ο Πρόεδρος, δεν είναι ερώτηση, είναι μια ε, παρότρινση. Να δώσετε την δέουσα προσοχή και στο θέμα του τουρισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Φιντάντσα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Υπουργέ, καλή τύχη. Θα επαναλάβω για τους προαλήσατε σε κάποια ζητήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η εργασία που έχει γίνει στο Κοινοβούλιο για τη δέσμη ειδικά με τα αεροδρόμια. Πάντα θέλαμε αυτοί οι τρεις κανονισμοί να ειδωθούν ως ένα πακέτο, μια δέσμη. Γνωρίζουμε ότι δύο εξ αυτών παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα από ότι ο τρίτος, αλλά θα πρέπει να κάνουμε θετικά βήματα προς την κατεύθυνση Λοιπόν, συμφωνώ σε εκ του με την έκκληση που έκαναν πολλοί συνάδελφοι, προκειμένου αυτό το θέμα να μην παραμείνει στα σιρτάρι. Ε, καταγράφω το γεγονό ότι συμπεριλάβατε τι προτεραιότητέ σα ε, και το ζήτημα του Clean Power for Transport, δηλαδή για την ανάπτυξη των υποδομών για τα ήταν ε, τα εναλλακτικά καύσιμα θα είναι κάτι το ιδιαίτερα επίπονο, ε, ιδιαίτερα σε επίπεδο Συμβουλίου, διότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι ο των μελών για τις ημερομηνίε θέσει εφαρμογή των νέων αυτών προβλέψεων, σε ό,τι φορά τη χρηματοδότηση και σε μια περίοδο ε, ισχυνών αγελάδων Υπάρχει και το λεπτό ζήτημα του ορισμού των ε, προτύπων, των ενίων προτύπων που ε, έχουν ε, μεγάλα βιομηχανικά συμφέροντα. Για τον τουρισμό εσείς αναφερθήκατε στο, στο φόρουμ του Βίλνιους τον Οκτώβριο ε, νομίζω ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλω για να μην καταλήξουμε στο να ανταλλάσσουμε καλές ιδέες που συχνά η μία είναι παρόμοια με την άλλη όπως τα διάφορα συνέδρια και εύχομαι πω με αυτή την περίπτωση να προκύψει κάποιο καινοτόμο μήνυμα προκειμένου να επιτευχθούν ε, θετικά βήματα για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Κύριο Μπένον για δύο λεπτά έχει το λόγο. Καλώς ήλθατε κύριε Υπουργέ. Εγώ θέλω να καλωσορίσω τα αρχικά σας σχόλια και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να αδράξετε αυτές τις προκλήσεις όπως κάνουμε και εμείς με το τέταρτο πακέτο για τα σιδηροδρομικά στην Επιτροπή μας. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου για την ανάπτυξη της ενίας αγοράς και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω και εδώ μιλώ ως σκιώδης εισηγητής για τα τεχνικά ζητήματα στο πακέτο αυτό Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην καθυστερήσουμε στην επεξεργασία του θέματος αυτού και συνεργαζόμαστε με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα για να καταλήξουμε σε κάποιο, κάποια κοινή θέση του Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε όμως να δούμε και από τη δική σας πλευρά, από την πλευρά του Συμβουλίου, να μην αφήσετε να χρονίσουν οι διαδικασίες και να καθυστερήσουν τα χρονοδιαγράμματα. Ξέρουμε ότι είναι διαφορετικό το σύστημα στι βαλτικέ χώρε, είναι διαφορετικό και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι ιδιαιτερότητε δεν θα καθυστερήσουν την έγκριση των θεμάτων αυτών και από την τεχνική πλευρά και σε ό,τι αφορά το άνοιγμα τη αγορά. Αν προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε μία πρόοδο στι δύο αυτέ κατευθύνσει, θα είναι θετικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε μοναχά τι τεχνικέ μεταλλαγέ και μετά να δούμε ότι δεν είναι ανοιχτέ οι αλλαγέ και δεν μπορούν τα τρένα να διασύζουν την Ευρώπη. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα σαν πακέτο. Επίση, αναφερθήκατε και στου ενιαίου εθέρε και πόσο έχει καθυστερήσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου που έχει εγκριθεί. Είναι πολλά τα οποία θα κερδίσουμε από την περάτωση του εγχειρήματο αυτού των ενιαίων εθέρων. Τέλο, για τον τουρισμό, νομίζω ότι έχουμε εδώ ένα ιδιαίτερο τομέα ε, τουρισμού που είναι ο ιστορικός τουρισμός, ο ιστορι... το τουρισμός ιστορικής κληρονομιάς. Έτσι μπορούμε να κάνουμε πιο ελκυστική την ε, Ευρώπη στον κόσμο και με την Ινδία και την Κίνα να γίνονται πιο πλούσιες χώρες, μπορούν έτσι να γίνουν πιο ελκυστικοί οι ευρωπαϊκοί χώροι, ιδίω από πολιτιστική άποψη. Δύο λεπτά, κύριο Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομο. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε για την ενημέρωση που δώσατε στην ε, Επιτροπή μα για τον ε, σχεδιασμό, τις προτεραιότητες και τους στόχους της Προεδρίας σας στον τομέα των μεταφορών που είναι ζωτικός για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Θα ήθελα να εστιάσω την παρέμβασή μου και τα ερωτήματά μου σε ένα θέμα. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πριν από μερικές εβδομάδες μια νέα πρόταση, πακέτο, για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Λιμένων, για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντίστοιχες απόπειρες για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας ευρωπαϊκής πολιτικής είχαν γίνει και στο παρελθόν, όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, χωρίς όμως να καταλήξουν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά ξεκινάει μια νέα σημαντική προσπάθεια. Θα ήθελα, εάν μπορείτε, να μας πείτε να μας δώσετε ένα γενικό σχόλιο, πώς βλέπετε αυτή την πρόταση, την πρώτη γενική σας αντίδραση και τι προτίθεστε και πώς προτίθεστε να χειριστείτε αυτό το τόσο κρίσιμο ε, ζήτημα και αυτή την πρωτοβουλία της Κομισιόν στο επόμενο σημαντικό εξάμεινο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Από τη δική μου πλευρά κύριε Υπουργέ θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στα εγχειρήματα αυτά που θα αναλάβετε ως πρόεδρος του Συμβουλίου και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ε, Λουθουανία. Από ό,τι ακούσατε υπάρχουν επαναλαμβανόμενα θέματα που έχετε πάρει συζήτηση, το τέταρτο συνδεδομικό πακέτο, η εφαρμογή για τους ανοιχτούς εθέρες, η προσπάθεια λοιπόν να μπορέσουν να προχωρήσουν όλα αυτά τα θέματα μέχρι το τέλος της ε, ε κοινοβουλευτικής περίοδου η βία Μπάλτικα είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εσάς μέσα στην ε, συνδυοδομική σύνδεση για τη Βαλτική, αλλά είναι και τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και φυσικά υπάρχει και το πακέτο για τα αεροδρόμια. Ξέρουμε το πρόβλημα με το πακέτο για τα αεροδρόμια είναι το προαιώνιο πρόβλημα των Ισπανών και των Βρετανών σε σχέση με τα αεροδρόμια στο Γιβραλτάρ, αλλά είπαμε και εμείς αφήστε το αυτό το καταραμένο το Γιβραλτάρ και ας προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα θέματα και εν καιρό θα μπορέσει να επιληθεί το θέμα αυτό ούτως ή άλλως από μόνο του. Δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε το Γιβραλτάρ να έχει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπειρο. Σας δίνω το λόγο λοιπόν κύριε Υπουργέ για να απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Μεταφορών, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που έσχον να ακούσω τα σχόλιά σας και να ακούσω το ενδιαφέρον το οποίο έχετε αναφέρει για τα θέματα αυτά. Πάνω από 10 μέλη της Επιτροπής σας έχουν λάβει το λόγο σχετικά. Αυτό καταδεικνύει ότι έχετε πολύ καλή γνώση των θεμάτων και είσαστε ιδιαίτερα έτοιμοι και πρόθυμοι να προχωρήσετε στην έγκριση αυτών των νομοθετικών πράξεων και να μπορέσει να αρχίσει έτσι η εφαρμογή αυτών των πράξεων. Δεν μπορώ να σας πω ότι νιώθω και πολύ άνετα ενώπιον σας, γιατί νιώθω το βάρος της ευθύνη. Είναι η πρώτη μας προεδρία ως Λιθουανία. Συγχρόνως όμως πιστεύω ότι αυτές οι προκλήσεις είναι και ευκαιρίες. Επομένως έχω ένα θετικό πνεύμα. Βλέπω ότι είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε μαζί μας. Γι' αυτό ελπίζω ότι η Λιθουανική Προεδρία θα είναι πράγματι μια επιτυχία. Θα ήταν δύσκολο για μένα να απαντήσω όλα τα ερωτήματά σας. Γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Απλώς θέλω να πω τα εξής όμως. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Νομίζω ότι η κύρια προτεραιότητα είναι να προωθήσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο και όχι των μεμονωμένων κρατών μελών. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την καλή θέληση που έχετε δείξει. Και θα ήθελα να σας πω ότι είναι φανερό ότι θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη η μέση διαταξή μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Η Λιθουανική Προεδρία δεν θα είναι μια εξάμηνη προεδρία, στην πραγματικότητα θα είναι 4,5 μήνες μονάχα. Έχουμε τις καλοκαιρινές διακοπές και μετά έχουμε <clears throat> το κενό διάστημα πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ είναι τεράστιος ο όγκος των θεμάτων που πρέπει να διεκπαιρέωσουμε. Ξέρετε, ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά θέματα που θα θέλετε να προσθέσετε στην ημερήσια διάταξη, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να παρατείνουμε το εξάμεινο της Προεδρίας. Δεν έχουμε αρκετούς πόρους, δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Και ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να βρούμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Αναφερθήκατε ιδιαίτερα στο τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα πολύπλοκο θέμα και ένα ευρύ θέμα. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή νομικούς, μερικά νομικά μερικά συγγνώμη, νομοθετήματα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε. Εγώ δεν είχα σαν στόχο να αναλύσω τις τεχνικές πτυχές αυτού του πακέτου ενώπιόν σας. Θέλω να περιοριστώ λοιπόν σε αυτά που σας λέω, ότι είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε όλα τα τεχνικά στοιχεία και να προχωρήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Προφανώς αυτές δεν μπορούν να είναι μεμονωμένες συζητήσεις, θα πρέπει να συνδέονται και με όλες τις άλλες πτυχές του θέματος. Άκουσα και κάποιες επικρίσεις σε σχέση με την διαμπάλτικα, ε, με την ε, σύνδεση της σιδεροδρομική. Υπήρξαν πολλές ε, ανησυχίες που διατυπώθηκαν και πολλοί, όπως ο κύριος Κράμερ, θα θέλαν να ξέρουν ποιο είναι το μέλλον αυτού του διαδρόμου, αυτού του εγχειρήματο για την σιδηροδρομική σύνδεση της Βαλτικής. Εδώ θέλω να πω ότι η χώρα μου αντιμετωπίζει το θέμα αυτό σαν δύο εγχειρήματα, δύο σχέδια. Το ένα έχει προχωρήσει κατά την απόψή μας με ικανοποιητικό τρόπο. Το 2015 θα έχουμε σιδηροδρόμους οι οποίοι θα συνδέουν ε, την Κάουνας με το, Ευρωπα... με το υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Δίκτυο και κύριε Κράμερ μπορείτε να έρθετε τώρα και να δείτε ότι θα κάνετε πολύ λιγότερο χρόνο. Το πρόβλημα είναι περισσότερο το Rail Baltica 2. Και εδώ εμπλέκονται και άλλα κράτη-μέλη, όχι μονάχα οι χώρες της Βαλτικής σε αυτό το εγχείρημα. Εάν δεν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, τότε τα βαλτικά κράτη θα παραμείνουν εναπομονώσει, δεν θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Η αρχή της αλληλεγγύης είναι πολύ σημαντική και επίσης είναι απαραίτητο να υλοποιήσουμε αυτό τον μεταφορικό ε, διάδρομο. Εγώ εκπροσωπώ την Ιλθουανική Προεδρία ενώπιό σα και πρέπει να πω ότι είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό για την Βαλτική. Ο στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις για το πώς θα μπορέσουν να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό οι στόχοι μας. Θέλουμε να βρούμε ένα νομικό εργαλείο για να κάνουμε πραγματικότητα όλα αυτά. Μπορεί να γίνει με μια κοινοπραξία. Μαζί με τη Λετωνία, την Εστονία, την Πολωνία, την Φιλανδία κτλ. Θα αναζητήσουμε εταίρους για να μπορέσουμε να κάνουμε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το εγχείρημα και φυσικά θα αναζητήσουμε και αλλού πόρους. Κατανοώ ότι, ότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι ο στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε πραγματικά αυτό το σχέδιο. Έχω μιλήσει και με τον αρμόδιο αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Σιμ Κάντας και έχει επίσης επικυρωθεί και από τον πρόεδρο της, την πρόεδρο της Λιθουανίας ότι θα γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά σε συζητήσει με άλλους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα αεροδρόμια τώρα να πω κάτι για το πακέτο για τα αεροδρόμια. Αναφερθήκατε στα θέματα αυτά που εμπλέκουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Όλα αυτά δεν θα, συζητήσουν, δεν θα σταματήσουν τις συζητήσεις μας και την αναζήτηση κοινού εδάφους. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν είχα χρόνο να απαντήσω όλα τα ερωτήματα συγκεκριμένα που θέσατε. Είναι χρήμα ο χρόνος. Ελπίζω ότι η συνεργασία μας θα είναι καρποφόρα και σας ευχαριστώ για, τις, για τα καλά σας λόγια. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Όπως είπα και στην αρχή, προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μαζί σας αλλά και με τους συναδέλφους σας ε, στο τμήμα μεταφορών του Υπουργείου σας. Το Κοινοβούλιο πάντα είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με την Προεδρία. Πάντα λέω στην εκάστοτε Προεδρία ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Ελάτε να μου μιλήσετε, να μου κάνετε προτάσεις, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη φυσικά της Επιτροπής. Ελπίζουμε ότι τον Ιανουάριο όταν θα έρθετε και θα μας μιλήσετε για τις επιτυχίες της Λιθουανικής Προεδρίας θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε και να σας χειροκροτήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Okay, guys, can we move on? Uh, those who need to... Κοιτάξτε, όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν, παρακαλώ πράξτε το ησύχως. Ε, το επόμενο θέμα στην μισεδίδαξη είναι το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο, αποτελέσματα και προοπτικές. Θα ακούσουμε παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πρόγραμματος Μάρκο Πόλο. Κύριος Καραμίτσης είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχα... το μέλη της Επιτροπής. Νομίζω πως έχετε κάποιο αντίγραφο της παρουσίασης. Οι οθόνες είναι πολύ μικρές για μένα, μόνο ότι φοράω γυαλιά. Εντάξει, λειτουργεί το σύστημα μεν, αλλά δεν μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Θα φροντίσω να το διατρέξω. Έχω 15 λεπτά στη διάθεσή μου και θα έχουμε και λίγο χρόνο για ερωταποκρίσεις. Θα είχαμε να κάνουμε μια ανακοίνωση, ότι αυτό απαιτείται από το άρθρο άρθρο του κανονισμού Μάρκο Πόλο. Δημοσιεύσαμε αυτή την ανακοίνωση στις 10 Μαρτίου 2013 και εστιάσαμε στα αποτελέσματα του προγράμματος και για την μετά το 2013 περίοδο, κάτι το οποίο συζητήθηκε ήδη όταν εξετάσαμε το νέο πλαίσιο. Επίσης υπήρξε και ένα έγγραφο ε, το οποίο περιλαμβάνει πολλά στατιστικά στοιχεία και απαντούσε σε μια σειρά από θέματα που αφορούσαν στο άρθρο 14 του κανονισμού του Μαρκοπόλου. Για τις επιπτώσεις του Μαρκοπόλου η εμπειρία από την ε, μεταφορά της διαχείρισης προγράμματος ε, στο ΕΑΣ και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο θέλω να τονίσω είναι το το σχεδιασμό του Μάρκο Πόλο. Έχουμε το Modal Shift. Επίσης έχουμε το χρηματοδότηση κινδύνου, τα αποτελέσματα του προγράμματος και το πιο χαρακτηριστικό είναι η λογοδοσία που υπάρχει για το πρόγραμμα αναφορικά με τα inputs και τα outputs. Και τι αυτό που είναι μοναδικό είναι ότι οι πληρωμές βασίζονται στις, ε, στο modal shift. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια σωστή ε, διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων. Το πρώτο πράγμα δίρκε σε τέσσερα χρόνια, από το 2003-2006, με τον προηγούμενο προβλησμό 102 εκατομμυρίων. Όλα τα, όλες οι βάσεις έχουν ολοκληρωθεί. Το δεύτερο πρόγραμμα ήταν από το 2007-2013. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά έχουμε 98 προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν το 2003 και 2012 και 55 από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί το Μάρκο Πόλο 1 και τα 143 εντάσσονται στο Μάρκο Πόλο 2 και ορισμένα εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπορούμε να σημειώσουμε πως πάνω από 700 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, περισσότερο εξ αυτών μικρομεσαίες, υποστηρίχθηκαν και εδώ βλέπετε την κατανομή των προγραμμάτων ανάμεσα στα χρόνια 2003-2012. Αναφέρομαι τώρα στα αποτελέσματα του Μάρκο Πόλο 1, όπου τα τελικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε το τι σημαίνει αυτό, σημαίνει 1230 φόρτιγα τα οποία κυκλοφόρησαν ανάμεσα στο Βερολίνο και το Παρίσι με ένα φορτίο 18 τόνων το, καθένα. Θα επανέλθω στο θέμα της δαπάνης των χρημάτων διότι δεν δαπανήθηκαν όλα τώρα για το Μάρκο Πόλο τα τελικά αποτελέσματα δεν είναι ακόμα διαθέσιμα. Το πρόγραμμα μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το 2019-2020. Το, το Model shift, η αλλαγή του μεταφοράς ε, αυξήθηκε μέχρι τώρα από σε 20 δισεκατομμύρια τόνα χιλιόμετρο Βλέπετε ότι έχει σχεδόν διπλασιαστεί η απόσταση σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα Μάρκο Δεν μιλάμε πια Παρίσι, απόσταση Παρίσι Βερολίνο, αλλά ε, Βαρσοβία Βουκουρέστη. Περισσότερα θα ε, επιτευχθούν ανάμεσα στο 2012-2013 και προσβλέπουμε σε μια διαφορά κατά 61 εκατομμύρια τόνους ανά χιλιόμετρο. Ή χιλιομετρικούς τόνους. Οι πληρωμές ε, στο πρόγραμμα ανέρχονται σε πάνω από 32 εκατομμύρια ευρώ για ένα σύνολο 41 τα οποία δαπανήθηκαν στο πρόγραμμα Μάρκο Πόλο 1 με βάση τον υπολογισμό που έγινε από την ΑΣΥ και εξωτερικούς συνεργάτες που το έλεγξαν, το εξωτερικό κόστος του Μάρκο Πόλο μπορεί να ανέλθει σε 432 εκατομμύρια ευρώ και προσβλέπουμε σε περαιτέρω ωφέλη από το πρόγραμμα αυτό. για κάθε ένα ευρώ που δαπανάμε έχουμε 13 που επιστρέφονται. Δηλαδή έχουμε έφερος 13. Τώρα για την χρήση του προπολογισμού, όπως σας είπα, ήταν χαμηλότερο, χαμηλότερη η επίδοση αυτό που πιστεύαμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι διατροπικές λύσεις είναι πιο περίπλοκες και δύσκολο να επιτευχθούν υπήρχαν προβλήματα διαλειτουργικότητας ε, σε φορά την διασύνδεση διαφορών τρόπων μεταφοράς και είχαμε μπει στην οικονομική κρίση, κατά τη της οποίας πολλοί δεν ήθελαν να αναλάβουν κανένα κίνδυνο και να αναλάβουν ε, να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις γιατί αυτό όμως έχει σημασία. Διότι δεν πετάξαμε τα χρήματα από το παράθυρο, πλούσαμε μόνο 42.000 από τα 102, εκατομμύρια από τα 102 που ήταν διαθέσιμα. Το 46% του στόχου επιτεύχθη, και τα 60 εκατομμύρια που δεν δαπανήθηκαν επιστράφηκαν στον προπολογισμό της Ένωσης. Για το Μάρκο Πόλο 2 πρόκειται για 75 εκατομμύρια τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Άλλα σημαντικά αποτελέσματα νομίζω θα πρέπει να υπογραμμίσουμε κάποια εξ αυτών. Πρώτα απ' όλα η αηφορία. Πολλά από τα προγράμματα συνεχίζουν μετά από το τέλος ε, της ε, περίοδου συμφωνίας χορήγησης ε, η αλλαγή του τρόπου μεταφορών θα ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερη από ότι αυτή που λεγόταν κατά την συμβατική περίοδο. Το ελάττωμα είναι ότι οι διαδικασίες είναι κάπως περίπλοκες, το μειονέκτημα μάλλον ε, αυτό. μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεώρησαν ότι το όλο σύστημα είναι κάπως περίπλοκο και δεν κατάφεραν να δαπανίσουν όλα τα χρήματα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο προτείναμε για το Μάρκο Πόλο 2 ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε βοηθητικές υποδομές Εάν αυτό ήταν δυνατόν, θα ήταν προ όφελο του προγράμματος, θα είχαμε μεγαλύτερη δυνατότητα δαπάνης κονδυλίων. Τώρα αυτό όμως ε, διορθώνεται στο σύμφωνα με το νέο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα κράτη-μέλη, ειδικά τα νησιωτικά, δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αυτό το μέσο. Ορισμένοι ανησυχούν για το ζήτημα του ανταγωνισμού μόνο ότι κάναμε πολλές ε, αναλύσεις δεν είδαμε ότι τελικά να προκύψει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τώρα τα επόμενα βήματα έχουμε μια νέα προσέγγιση και ε, έχουμε συναγάγει κάποια διδάγματα από το από τα προγράμματα του Μάρκο Πόλο, το, το πλαίσιο πολιτικής, ε, τα Trans-European Transport Network Program, ε, έχουμε άλλα θέματα που αφορούν ε, τις τους σιδεοδρόμους, τις θαλάσσιες μεταφορές για τις σχετικές υποδομές. Θέλουμε επίση να διευκολύνουμε τις ε, διατροπικές ε, μεταφορές Κοιτάξαμε φυσικά και τη νέα πλευρά της, ε, κάποιες πλευρές της καινοτομίας. Όλα φυσικά δεν σημαίνουν ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι τρόποι μεταφορών, αλλά οι νέες καινοτομίες σίγουρα μπορούν να τύχουν στήριξη από το πρόγραμμα. Επίσης προσπαθούμε να δούμε πώς ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες ελλείψεις ε, που προκύπτουν στις αγορές. Δεν έχουμε φτάσει στον τελικό, προσδιορισμό των υπηρεσιών Μαρκο ε, Πόλο. Θα υπάρξει μια εξάντε λεπτομερή ανάλυση για το σύμφωνα με το 38 αλλά θα λάβουμε υπόψη φυσικά τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες που προέκυψαν από το πρόγραμμα και αναβίβολα θα έχουμε ένα σημαντικό όφελος από όλα αυτά για τα προσεχή αυτά που τον παρόν πρόεδρε. Νομίζω ότι λάβατε ήδη και την ανακοίνωση και το σχετικό έγγραφο. Είμαι έτοιμο να απαντήσω σε ερωτήσεις και σχόλια το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Γκρόσο, ο κύριος Αλκατρό η κυρία Μάιζερ από το λόγο. Κάποιος άλλος δεν λάβει το λόγο. Ο κύριος Κόλιτσεκ. Άλλος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάποια σχόλια και κάποιες παρατηρήσεις. Για μας το Μάρκο Πόλο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό πρόγραμμα και ανταποκρίνεται σε πολλές ε, προσδοκίες να έχουμε καλύτερη τροπική κατανομή των ε, μέσων μεταφοράς. Τι κάνετε όμως για να μπορέσετε να ξεπεράσετε την πολυπλοκότητα που είδατε στο πρώτο στάδιο αυτού του εγχείρηματος. Πιστεύω ότι αν δείτε τόσο μεγάλες δυσκολίες θα πρέπει να τροποποιήσετε την ε, μέθοδο που θα ακολουθήσετε και δεν μπορούν να αποτυγχάνουν τα προγράμματα αυτά λόγω της πολυπλοκότητας. και θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει και κάποια καλύτερη παρακολούθηση του εγχειρήματο αυτού. Για μένα από θεσμική άποψη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αν θέλουμε σιγά σιγά να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, ιδίως τα θέματα τα οποία είναι τόσο πολύπλοκα. Ο κ. Αλχανταράουι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με την ερώτηση. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την γεωγραφική κατανομή. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου αυτού του είδους τα προγράμματα χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις άλλες χώρες. Και σε σχέση με αυτό έχετε την αίσθηση ότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο Είναι γνωστές οι ευκαιρίες που προσφέρει. Το γνωρίζουν όλες οι επιχειρήσεις, δηλαδή τι μέσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το μέλλον. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε για τις αμφιβολίες που υπάρχουν σε σχέση με τον προπολογισμό. Δεν μπορούμε όμως να ξέρουμε περισσότερα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αν μη τι άλλον σχετικά με την προκήρυξη, κάτι σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, πώς θα προχωρήσει. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καραμίτσο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία Εγώ θέλω να επαναλάβω κάποια ερωτήματα που τέθηκαν. Ποια είναι η κατανομή των εγχειρημάτων σε διάφορα κράτη-μέλη και μπορεί πράγματι να υπάρξει αυτή η μετακίνηση από τα φορτηγά, ένα εκατομμύριο φορτηγά να μεταφερθούν σε εσωτερικούς υδάτινους δρόμους και σε σιδηροδρόμους και μπορείτε επίσης μέσα από τα προγράμματα του Connecting Europe να εξασφαλίσετε και, με μεγαλύτερη, και μεγαλύτερη μεταφορά στους εσωτερικούς υδάτινους ε, δρόμους της Ευρώπης. Αυτό θα με ενδιαφέρει να ξέρω. Ο κύριος Κράμερ. Κρίμα που αυτή η αντιμετώπιση δεν έχει καρποφορήσει γιατί στην αρχή η, τα κίνητρα τα οποία είχαν θεσπιστεί είχαν και σύνδεση με την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Όποιος δηλαδή μεταφέρει από το δρόμο στα, στους εσωτερικούς υδάτινους δρόμους στο σιδηρόδρομο παίρνει κάποιο κίνητρο γιατί αντιμετωπίζει και την κλιματική αλλαγή. Αλλά τώρα εφόσον είδαμε αυτές τις ελλείψεις το θέμα είναι πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα μεταφερθούν τώρα όλα αυτά τα πράγματα στο Connecting Europe στη διευκόλυνση αυτή. Αν υπάρχει λοιπόν η σχεδίαση αυτή, δεν ξέρουμε αν θα, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο ξεκινάει και προχωράει και ακόμα και αν δεν έχει υπερατωθεί, ξαφνικά κλείνουμε τη στρόφιγγα και σταματάει η χρηματοδότηση. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το σύστημα εμπορία εκπομπών. Αυτό είναι ένα νέο σύστημα, θέλουμε να το προωτήσουμε. Υπήρξαν σφάλματα στην αρχή, έχουμε εκδώσει πάρα πολλά πιστοποιητικά ε, για εκπομπή αριών θερμοκηπίου. Έχει πέσει σαν συνέπεια η τιμή του και έχει καταρρεύσει η αγορά, αλλά πρέπει να υπάρξει εδώ μια βελτίωση. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει προσπάθειες, αλλά τονίζουμε ότι αυτό ήταν ένα θετικό εργαλείο. Απλώς κάναμε λάθη στην εφαρμογή αυτού του εργαλείου. Γιατί, γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν δεν προβαίνει σε μια ανάλυση και εξετάζει τις ελλείψεις, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να υπάρχουν κίνητρα όταν μειώνονται οι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Αυτά τα έχει απεμπολίσει η Κομισιόν. Έχει φύγει λοιπόν από τους στόχους για την κλιματική αλλαγή. Γιατί? Γιατί μέσα στην ε, Connecting Europe, στο διευκόλυνση αυτή, δεν έχετε κανένα απολύτως κριτήριο. Αδιακρίτως χρηματοδοτείτε όπου μπαίνει τσιμέντο και φτιάνετε κάτι καινούριο. Αυτή λοιπόν η καλή ιδέα που είχατε στην αρχή, τα συνδέετε αυτά με την κλιματική αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, αυτά τα έχετε καταργήσει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ποια είναι η θέση της Κομισιόν σχετικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριο Σκόλτσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Να μην επαναλάβω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Αυτό όμω που θέλω να συμπληρώσω είναι μια ακόμα ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε ποιοι είναι οι τομείς που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο. Θέλω δηλαδή κάποια παραδείγματα. Πριν από 20 περίπου χρόνια ξαναφτιάξαμε ένα εργοστάσιο το οποίο κατασκεύαζε διάφορα προϊόντα από γυαλί. Και μάθαμε ότι τα αντικείμενα αυτά δεν μεταφέρονται πια δια γιατί αξίζει μόνο λέει άμα είναι πάνω από 800 χιλιόμετρα η απόσταση. Αλλιώς ε, δεν αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιείται το τρένο. Να λοιπόν ένα παράδειγμα μιας μεγάλης βιομηχανικής παραγωγής, αλλά λέγανε ότι κάτω από 800 χιλιόμετρα δεν άξιζε τον κόπο. Λοιπόν, εσείς τι λέτε, υπάρχει ένας τρόπος να αξίζει τον κόπο, γιατί πρέπει να μπορεί να είναι χρήσιμο. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορεί να ακουστώ γελίο, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θέλω να ικανοποιήσω την περιέργειά μου. Θέλω να μάθω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να μα περιγράψει μία δραστηριότητα έτσι κλασική Μάρκο Πόλο, τυπική, χαρακτηριστική. Μπορεί να μα περιγράψει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση Μάρκο Πόλο για να καταλάβουμε καλύτερα πώ λειτουργεί. Γιατί τη γενική ιδέα την αντιλαμβάνομαι, αλλά θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριμένο, ένα παράδειγμα δηλαδή να μας δώσει. Πρόεδρος. Κύριε Καραμίτσο. Ναι, εγώ ξέρω γιατί το ονομάζουμε Μάρκο Πόλο, ξέρω πώς είναι το έμβλημα, τέλος πάντων. Εγώ το κατανόμασα εξάλλου. Λοιπόν, παρακαλώ, εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για τις πολυάριθμες ερωτήσεις και σχόλιά σας. Κοιτάξτε, δεν θέλω να προκαταλάβω βέβαια την ε, έκθεση του λεγκτικού συνεδρίου, οπότε προσπαθώ να μην ε, πω υπερβολικά πολλά για το πρόγραμμα πριν δω την έκθεση αυτή, γιατί να ξέρετε ότι έχουμε πετύχει πολλά από αυτά που θέλαμε να πετύχουμε και το μόνο που μας δυσκόλεψε ήταν οι διοικητικοί κανόνες που επιβάλλουμε στις επιχειρήσεις. Ήταν ο δημοσιονομικός κανονισμός δηλαδή, ο οποίος έπρεπε να εφαρμοστεί. Αλλιώς, κατά τα άλλα, θα έλεγα, προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα, πήραμε τα μαθήματά μας από το πρόγραμμα Μάρκος Πόλος 1, να ξέρετε ότι άρχισε μεγαλύτερη διαφήμιση. Έχουμε, θα έλεγα, προγράμματα κυρίως μεταφοράς προς τους σιδηρόδρομους και τις θαλάσσιες μεταφορές. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες μεταφορές και μέσω πλωτών ε, υδάτινων διαδρομών δηλαδή στην εδώ Ένα πάντως από τα προβλήματα που έχουμε είναι η δομή της βιομηχανίας, γιατί πρόκειται για μικροεπιχειρήσεις, δεν είναι καν μεσαίου μεγέθους, είναι μικρές επιχειρήσεις με έναν ίσως. Οπότε οι επιχειρήσεις που έχουν 10-15 πλοία θα μπορούσαν να διαφερθούν περισσότερο για το πρόγραμμα και να συμπεριληφθούν στα προγράμματά μας. Αλλά αν δείτε τα προγράμματά μας δεν υπάρχει καμία επιχείρηση με ένα μικρό πλοίο που να προσπαθεί να επωφεληθεί και να μεταφέρει έτσι τα εμπορεύματά της. Έχουμε περισσότερες επίσης επιχειρήσεις που μας έρχονται ως ε, ομάδα. Εξαιτίας της διαφήμισης ίσως που γίνεται, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Έρχομαι τώρα στις ερωτήσεις. Κύριε Ρικέ, που θέλετε παραδείγματα. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. δικές μεταφορές μεταξύ βορειοδυτικής Γερμανίας και Βόρειας Ισπανίας. Εδώ έχουμε προγράμματα τα οποία έχουν καταφέρει να απομακρύνουν από τους δρόμους τα φορτηγά και μέσω θαλάσσης να κάνουν τη μεταφορά. Επίσης πολλά αστυνομικά προγράμματα υπάρχουν που εξυπηρετούν για παράδειγμα Πολωνία με Βόρεια Ιταλία. Αντί δηλαδή τα φορτηγά να πηγαίνουν από το δρόμο, από τον αυτοκινητόδρομο, τα φορτώνουν τα εμπορεύματα στους σιδηροδρόμους, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής. Γεωγραφική κατανομή. Καλή ερώτηση. Και ίσως θα έπρεπε να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε, ίσως να σας στείλουμε τα διάφορα προγράμματα, ώστε να δείτε εσείς καλύτερα γεωγραφικά πώς γίνεται η κατανομή. Πάντως με εξαίρεση κάποιες απομακρυσμένες περιοχές Μάλτα, Κύπρος, τέτοια μέρη ακόμα και την Ιρλανδία, που έχουν χρησιμοποιήσει καλά το πρόγραμμα, θα έλεγα ότι για τις υπόλοιπες η γεωγραφική κατανομή είναι αρκετά ισόρροπη. Τώρα για την πολυπλοκότητα. Πολύ σωστά το λέει ο κύριος Γκρός και πώς θα αλλάξουμε τις διαδικασίες. Προσπαθούμε να τις απλοποιήσουμε από το Μάρκο Πόλο 1 στο 2, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει τόσο όσο θα θέλαμε. Τώρα με τη νέα προσέγγιση που θέλουμε να ακολουθήσουμε με την εξάντια ανάλυση που κάνουμε για τις υπηρεσίες στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2016 και τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα, παίρνουμε μαθήματα από το παρελθόν για τα αδύναμα σημεία και ελπίζουμε να πετύχουμε την απλοποίηση. Μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε είναι εξή. Πολλέ επιχειρήσει που θέλανε να, να συμμετάσχουν θέλανε να καλυφθεί το τελευταίο χιλιόμετρο. Να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση σε κάποιο τέρμιναλ ή να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν ε, την ε, ε, μεταφορά του τελευταίου χιλιόμετρου. Κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό με το Μάρκο Πόλο 1. Τώρα δεν ξέρω ο κύριος Κουμτσάκος, α δεν είναι πια εδώ. Καλά, είναι άλλοι όμως οι συζητητές στα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα νομίζω ότι είναι εφικτό αυτό πια. Οπότε θα υπάρξει βελτίωση στο μέλλον. Για το μέγεθος των προγραμμάτων τώρα. Πράγματι, δεν είναι πολύ μεγάλα τα προγράμματα. Τα περισσότερα είναι για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρά προγράμματα με καλά αποτελέσματα όμως. Για τον κύριο Κράμερ και την προστασία του περιβάλλοντος ομολογώ ότι δεν κατάλαβα πολύ καλά τι εννοείται. Αλλά είναι σαφές ότι το πρόγραμμα αυτό έχει την περιβαλλοντική διάσταση. Αποτελεί στοιχείο κλειδί για το αποτέλεσμα. Για ένα ευρώ που ξοδεύουμε θέλουμε 13 ευρώ περιβαλλοντικό αποτέλεσμα είτε πρόκειται για την ηχορύπανση, είτε πρόκειται για τις εκπομπές ε, ρήπων κλπ. Είναι σαφές, έχει υπολογιστεί. Και είναι ένα θετικό στοιχείο αυτού του είδους ε, δράσης. Όταν δηλαδή μεταφέρονται τα εμπορεύματα με άλλους τρόπους μεταφοράς πέρα των οδικών. Τα περιβαλλοντικά κέρδη δηλαδή υπάρχουν το ξέρουμε, έχουν αποδειχτεί. Τι άλλο, νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Α, τι είδο εμπορεύματα. Χαλιβουργία, έπιπλα, τρόφιμα, μεταφέρονται. Αυτά είναι τα κύρια εμπορεύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Εκτός μικροφώνου μια παρέμβαση του κύριου Κράμερ. Και πώς το κάνετε αυτό με τα κίνητρα. Νομίζω ότι αυτό το συζητήσατε πάντα ο κύριος στη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά δίκτυα όταν συζητήσατε για τις εμπορικές υπηρεσίες. Ένα από τα στοιχεία περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση, τα περιβαλλοντικά ωφέλη δηλαδή. Καινοτομία, μεταφορά αγαθών, περιβαλλοντικά ωφέλη είναι μέσα στο άρθρο 38. Είναι όμως πολύ νωρίς τώρα για να πούμε σε τι βαθμό. Αλλά προς το παρόν αυτά τα μαθήματα έχουμε πάρει, αυτά σας παρουσιάζω σήμερα. Και τα αποτελέσματα τα χρησιμοποιούμε όσο γίνεται καλύτερα για να προχωρήσουμε σε παρετέρω βελτιώσεις. Σαϊντ. Ναι, και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το θέμα του ΣΕΦ για το μέλλον. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Η προκήρυξη διαγωνισμού, οι νέες προτάσεις, πώς θα οργανωθούν. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε περισσότερο, το χρονοδιάγραμμα δηλαδή. Στο ΣΕΦ υποθέτουμε ότι οι περισσότερες χώρες μέλη θα υποβάλουν προτάσεις, ενώ το Μάρκο Πόλο έχει να κάνει περισσότερο με ιδιωτικέ μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπατε. αυτά τα μικρότερα προγράμματα, τι επεξεργασίες θα τύχουν μέσω του ΣΕΦ. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Το άρθρο 38 για τις εμπορικές υπηρεσίες δεν λέει ότι μόνο οι χώρες μέλη μπορούν να υποβάλουν πρόταση. περιμένουμε στο δεύτερο εξάμεινο του 2014 μετά την εξάντη αξιολόγηση να έχουμε τις πρώτες προτάσεις για να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Άρα ήδη σε αυτήν την θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε προτάσεις για αυτού του είδους δράσεις βάσω του άρθρου 38 των ΤΕΝΤΗ με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα ευρωπαϊκά δίκτυα και το ΣΕΦ. Έχουμε ξεκινήσει την εξάντια αξιολόγηση για αυτού του είδους δράσεις βάσει του άρθρου 38, οπότε αρχές της επόμενης χρονιάς θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα του τι θα καλύψουμε με τις πρώτες προτάσεις, τα μέσα της χρονιάς δηλαδή. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Πρόεδρος. Καλώς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καραμίτσο. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ήτρε για το ΚΑΡΣ 2020. Εισηγητής είναι ο κύριος Βλασάκ. Παρακαλώ κύριε Βλασάκ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Και τώρα να σας κάνω εισαγωγή σε αυτή την ε, πολύ σημαντική νομοδότηση που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλής και που αφορά στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και την σταθερότητα. Γνωρίζετε πως βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη και σκληρή και είναι η πέμπτη συνεπτή χρονιά που η αυτοκινητομηχανία αντιμετωπίζει προβλήματα και αυτό αφορά πολλές ε, επιχειρήσεις ε, διότι τις αναγκάζει να αναδιαρθώθουν ορισμένες εξ αυτών χρειάζεται να σταματήσουν την παραγωγή τους. Δεδομένου του ότι αυτό αφορά 12 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης ε, άμεσα ή έμεσα, καταλαβαίνετε ότι ο κλάδος έχει ιδιαίτερη σημασία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα πρόγραμμα δράσης ώστε να μπορέσει η αυτοκινομηχανία να, ξεφυ... να βγει από το αδιέξοδο. Δεν θα ήθελα να αναφέρω εδώ όλες τις λεπτομέρειες, αλλά πρόκειται για τέσσερις άξονες, τέσσερις βασικούς άξονες. πρέπει να κατανοήσουμε ότι καθένας από αυτούς τους στόχους στηρίζονται σε μια στρατηγική που δεν είναι πάντα σαφής και ξεκάθαρη γιατί η Κομισιόν ε, προτείνει κάποιες ε, νομοθετικές πράξεις κατακαιρματισμένες προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Το βασικό πρόβλημα είναι πως η Ευρωπαϊκή Τροπή προετοιμάζοντας το πρόγραμμα δράσης φαίνεται πως ε, ανέπτυξε ένα σενάριο πολύ πιο αισιόδοξο από αυτό το οποίο πράγματι ισχύει στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε από 17 εκατομμύρια το 96 σε 11 εκατομμύρια χρειάζεται ως εκ τούτου να γίνουν αναδιαρθρώσεις ε, και σε αυτό το επίπεδο παραγωγής η κατάσταση έχει δημιουργήσει όπως καταλαβαίνετε πολλές δυσκολίες. Χρειάζεται να θέσουμε ορισμένες προτεραιότητες για αυτόν τον κλάδο ε, αυτή τη μηχανία βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις είναι αρνητικές, η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά, ως εκ τούτου χρειάζεται να αποταθούν λύσεις μια συγκεκριμενοποίηση προγράμματος δράσης. Ε, για τον λόγο αυτό χρειάζεται συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας ε, υψηλού επίπεδου με την οικονομία CARS 2002, 2020 και τρίτον χρειάζεται να ξεκινήσει μια μελέτη έτσι ώστε να δούμε την να κάνουμε μια μελέτη αξιολόγησης ε, αντικτύπου. Δεν χρειάζεται να αφήσουμε άλλο χρόνο να κυλήσει. Πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την αυτοκινητομηχανία και για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να παρεύουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν οι παραγωγοί να πετύχουν στόχους του περιβαλλοντικού ή άλλους. Είμαι πεπισμένο ότι αν αναγκάσουμε τους παραγωγούς να ε, ασχοληθούν με θέματα αεροδυναμικής κλπ. μπορούν νέες, νέες δυνατότητες ε, να προσφέρουν πολλά. Υπάρχουν και άλλα ζήτημα όπω οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, τα καύσιμα αλλά και τα ελαστικά. Εάν μπορέσουν οι βιομηχανίες να επιλέξουν κλάδους, τότε σίγουρα θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Πρέπει επίσης ε, να βελτιωθούν οι υποδομές σε πολλές χώρες ε, και δεν μιλάω μόνο για δρόμους αλλά και την υποδομή για, την, για τα ελεκτικά καύσιμα. Περιμένω τα ε, σχόλιά διότι ο κλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για τον αριθμό θέσεων απασχόλησης αλλά και για την έρευνα και την καινοτομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Φέρμπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έξω ονόματος του ΕΛΚ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό για την ανάπτυξη της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας να υπάρχει μια σωστή θέση της Επιτροπής Μεταφορών γενικά θέλουμε εμείς να τονίσουμε ως Επιτροπή Μεταφορών την δυνατότητα να προωθήσουμε τις εναλλακτικές μεθόδους αυτοκίνησης, τεχνολογίες αυτοκίνησης και αυτό απαιτελεί και γι' αυτό που αποτελεί προϋπόθεση να υπάρξει και καλύτερη εναρμόνιση στον τομέα αυτό Πρέπει να υπάρξει λοιπόν κάποια πρόοδος, θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινά πρότυπα για την ηλεκτροκίνηση μαζί και με τους Αμερικανούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα τρίτο στοιχείο, όπως ελέγχθη, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές. Δεν φτάνει να έχουμε εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτικέ μεθόδου κίνηση. Θα πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητε υποδομέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αυτέ οι αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα ή εναλλακτικέ πηγές κίνησης και νομίζω ότι κατά τα άλλα συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά τα οποία λέει ο εισηγητής. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή γνωμοδότηση που μπορούμε να δώσουμε στην Επιτροπή Βιομηχανίας για να τονίσουμε αυτά που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκάλια Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εν μεγάλη συντομία εξ ονόματος των σοσιαλιστών θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα σχόλια που μας έδωσε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να χαρούμε για το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει διατυπώσει αυτή την πρόταση γιατί σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι είναι μια σωστή πρόταση και κυρίως μια αναγκαία πρόταση όλοι μας συμμεριζόμαστε στην Επιτροπή Μεταφορών όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στρατηγική σημασία που έχει η αυτοκινητοβιομηχανία μέσα στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό ιστό και γι' αυτό πρέπει να διαμορφώσουμε όλου του απαραίτητου μηχανισμού ώστε αυτό ο τομέα να εξακολουθήσει να είναι ισχυρό και ανταγωνιστικό και φυσικά και βιώσιμο. Αυτό είναι και ο στόχο τη πρόταση τη Κομισιόν και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ηγετική θέση που έχει κρατήσει η Ευρώπη σε όλο τον κόσμο στην αυτοκινητοβιομηχανία, γεγονό ότι τα στοιχεία για τι πωλήσει αυτοκινήτων στην Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα θετικά και είναι σε κάμψη ο τομέα αυτό. Επομένω, απαιτεί μια αποφασιστική <clears throat> υποστήριξη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα άλλα θεσμικά όργανα. Λοιπόν, συμφωνούμε σε όλα αυτά τα σημεία με τον εισηγητή. Υπάρχουν άλλα σημεία στα οποία έχουμε κάποιε αποχρώσει να διατυπώσουμε. Όπως ε, είπα, το σχέδιο αυτό θα πρέπει να τεθεί το ταχύτερο δυνατόν σε εφαρμογή, να κάνουμε σαφή όλα τα μέτρα τα οποία θέλουμε να θέσουμε σε κίνηση και ποια είναι τα εργαλεία τα οποία θα υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο. Έχω όμως τώρα ορισμένες διαφοροποιήσεις. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια παρεξήγηση ή αν είναι διαφορετική η θέση μας. Παραδείγματος χάρη για τους στόχους σε ό,τι αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Εδώ η άποψή μας, η οποία... Η άποψή η οποία θα μεταφερθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει καταφέρει να επιτύχει μια συνολική συμφωνία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε εμείς να ανατρέψουμε αυτή τη συμφωνία τουλάχιστον μέχρι να δούμε ποια είναι η συνολική συμφωνία που θα επιτευχθεί μεταξύ Επιτροπή Περιβάλλοντο και Συμβουλίου, γιατί η Επιτροπή Περιβάλλοντο εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προφανώ συνεργάζεται με την αυτοκίνητο βιομηχανία, έχει δώσει δανειοδοτήσει, εγγυήσει δανείων για να μπορέσει η αυτοκίνητο βιομηχανία να προχωρήσει περισσότερο στην καινοτομία και στην έρευνα και να έχει μεγαλύτερη ευκαι... περισσότερες ευκολίες για να χρηματοδοτήσει αυτές τις ενέργειες καινοτομίες. Και εδώ Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήδη υπάρχει δράση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζες Επενδύσεων και αυτό ισχύει επίσης και με την ομάδα υψηλού επίπεδου. Δηλαδή η ανακοίνωση της Κομισιόν ήδη βασίζεται στην προηγούμενη επεξεργασία της ομάδας υψηλού επίπεδου και επομένως πρέπει να ενισχύσουμε το έργο της ομάδας υψηλού επίπεδου και τη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για να καθορίσουμε καλύτερα τις προτεραιότητές μας. Εν πάση περιπτώσει όλοι συμφωνούμε για τις γενικές γραμμές, δηλαδή ότι θα πρέπει να θέσουμε στην διάθεση της βιομηχανίας αυτοκίνητων όλα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από τις πολιτικές που θα αποφασιστούν από εμά, γιατί πρόκειται για ένα ιδιαίτερα στρατηγικό τομέα και δεν πρέπει να χάσουμε το τρένο της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ανταγωνιστικότητας με, αν δεν δράσουμε εγκαίρως. Κύριε Γκρίσμπεκ. Ευχαριστώ. Τα ίδια πιστεύω κι εγώ. Δεν ε, πρέπει να δυσκολέψουμε την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης που περνάει από τη χειρότερη κρίση της ιστορίας της. Πρέπει να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Καθημερινά ακούμε άσχημα νέα. Γι' αυτό ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ε, έκθεση για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βρούμε λύσεις ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να αποκτήσει νέα δυναμική. Αν εγκαταλείψουμε την ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία είναι σαν να εγκαταλείπουμε την ε, βιομηχανία στην Ήπειρό μας. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι από την έκθεση Βλασάκ πρέπει να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες που να προχωρήσουν με διαβούλευση όπως όλοι χαιρετίζω και εγώ το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης που προβλέπει τέτοιες συγκεκριμένες δράσεις και που θα μπορούσε να συμπληρωθεί, να διευκρινιστεί σε διάφορα σημεία. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Φέρμπερ. Έτσι, η ανανέωση της ευρωπαϊκής αυτοβιομηχανίας θα εγγραφεί στα πλαίσια της στήριξης που δίνει σε βιομηχανίες κλειδί η Ευρώπη όπως είναι αυτός που πρέπει βέβαια να προσαρμοστεί στις σημερινές προκλήσεις. Είναι θλιβερό να διαπιστώνουμε ότι ακόμα δεν έχουμε ένα πραγματικά ηλεκτρικό αυτοκίνητο που να έχει ευρωπαϊκό όνομα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και να προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία στα πλαίσια των πολιτικών μας. Γιατί να μην αναπτύξουμε μεγάλα προγράμματα με ενισχυμένη συνεργασία, να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας, ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε πρωταθλητές στην βιομηχανική έρευνα εδώ στην Ευρώπη. Γιατί να μην προβλέψουμε, για παράδειγμα, η Ευρώπη είναι ο πρωταθλητής των καθαρών μεταφορών. Εννοείται ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται συνεργασία και διαβούλευση. Και για να μην μακρηγορήσω, τρίτο σημείο μου. Δεν μπορεί να υπάρξει τεχνολογική καινοτομία αν δεν πρικοδοτηθεί και ανάλογα. Γι' αυτό καταδικάζω και εγώ το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει πετύχει το 3% του έπτης να το δίνει στην έρευνα και την ανάπτυξη. Χρειάζεται συγχρόνως οι τράπεζες να δανείζουν επαρκώς, να προσφέρουν δηλαδή πιστώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε φτιάξει ένα ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση για να βοηθήσουμε εκείνους που απολύονται από τη βιομηχανία και βρίσκονται στην ανεργία. Όντως, οι μισθωτοί αυτοί είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης. Γι' αυτό και εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο με την διαβίου κατάρτιση, ώστε οι μισθωτοί αυτοί να προσαρμόζονται και αν χάσουν τη δουλειά τους να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε άλλους τομείς. Αυτές είναι κάποιες πρώτες σκέψεις για την έκθεση του συναδέρφου. Και εννοείται ότι με όλους τους συναδέρφους και την κυρία Μάσινα και άλλους θα υποβάλουμε τροπολογίες για να μπορέσουν να περάσουν οι θέσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόλτσεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, έχω κάποιες παρατηρήσεις παρακαλώ. Γιατί βλέπετε δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για αυτό το θέμα. Θέλω να επιμείνω στο εξής. Για το 2020 ο αριθμός ή μάλλον τα περισσότερα οχήματα που θα έχουμε θα κυκλοφορούν με παραδοσιακά καύσιμα, με βενζίνη. Ίσως θα έπρεπε να δούμε τι στήριξη μπορούμε εμείς να δώσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανακύκλωση των οχημάτων αυτών και να προσπαθήσουμε να επεξεργόμαστε καλύτερα τα καύσιμα. Αυτοί είναι παράγοντες που είναι αναγκαίοι για να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα καύσιμα. για τα παραδοσιακά οχήματα, τα συμβατικά, αυτά θα εξακολουθούν να κυριαρχούν στο τοπίο. Πρέπει συνεπώς να έχουμε και άλλους στόχους για άλλου τύπου οχήματα και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλες αναλλακτικές πηγές ενέργειας, μπαταρίες για παράδειγμα που να μπορούμε να τις φορτίζουμε γρήγορα και εύκολα όπως τα ηλεκτρικά οχήματα. Και πρέπει να τυποποιηθεί ολόκληρος εξοπλισμός. Αυτό θα ήταν καλό να γίνει έγκαιρα εκ των προτέρων. Επίσης, θα έπρεπε να έχουμε και βρυδικά οχήματα για να μπορούμε πιο εύκολα να περνάμε από τα παραδοσιακά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια. Τα ευρυδικά οχήματα πιστεύω ότι είναι πολυβολικά στην πράξη. Τα ηλεκτρικά οχήματα φυσικά και είναι κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κάποιος να βάζει και στην πρίζα. Άρα χρειάζεται ανάπτυξη σχετικών υποδομών για να μπορούν τα οχήματα αυτά να φορτίζονται εύκολα. Πρέπει οι στόχοι αυτοί να προχωρήσουν ρεαλιστικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουν. Ευχαριστώ τον κύριο Κόλιτσεκ, λέει κύριος <clears throat> Κουν, γιατί αντιμετώπισε ήδη τα τεχνικά ζητήματα και αυτά συνδέονται με την ε, έρευνα και την ανάπτυξη νέων κινητήρων. Έχουμε ήδη θεσπίσει μια σειρά από για το περιβάλλον σε ό,τι αφορά την ε, ρήπανση, από διοξίδιο του άνθρακος και οξίδια του αζότου μέχρι το 2020. Και μιλάμε για το αυτοκίνητο που θα εκπέμπει 95 γραμμάρια το χιλιόμετρο διοξιδίου του άνθρακος. Αλλά τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Τι μορφή αυτοκίνητα θα έχουν αυτά. Θα πρέπει να ξέρουμε τι προκύπτει από την καύση ενός λίτρου δίζελ είναι 2,9 χιλιόμετρα. Μετά βλέπετε πόση απόσταση μπορεί να κάνει και επομένως μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι εκπομπές που θα πρέπει να έχουμε το 2020. Θέλουμε να έχουμε αυτοκίνητα που θα καίνε 3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. ακόμα και στους λομπίστες θα πρέπει να θέτουμε αυτό το ερώτημα. Ξέρετε τι τεχνικές θέλετε να προωθήσετε. Αυτό είναι μία πλευρά μονάχα. Το άλλο θέμα είναι η ενεργειακή απόδοση των κινητήρων και για τα φορτηγά και για τα ιδιωτικά επιχειρήματα, ε, ε, ε, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το να χρησιμοποιήσουμε και την ενέργεια του φρεναρίσματος και να τη χρησιμοποιήσουμε ως ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε πιο πολύ καιρό για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα όταν μιλάμε για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας σε ηλεκτρική μορφή που προκύπτει από την μη χρησιμοποιημένη ισχύ του κινητήρα. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά, πώς μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε. Οι, ιοντικές μπαταρίες λιθίου. Αν πρέπει να μεταφέρει κανείς το βάρος αυτών των ε, συσσωρευτών, τότε δεν έχει νόημα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μια βελτίωση στους τρόπους ε, αποθήκευσης της ε, ενέργειας σε μπαταρίες ιόντων λιθίου. Ο κύριος Κόλτσεκ μίλησε για τους κινητήρες υδρογόνου και κυψελών καύσης και αυτή τη μορφή θα πρέπει να προωθήσουμε για κίνηση οχημάτων και γι' αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δώσουμε και μια σύνδεση με τον ορίζοντα 2020 το μόνο το οποίο μπορώ να υποστηρίξω είναι ότι σπαταλάμε απίστευτες πορεί, ποσότητες ενέργειας. Δεν είναι θέμα οπισθοφόρτησης και επιστοποιητικών για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Λένε ότι, λέμε ότι πρέπει να κάνουμε πιο ακριβά τα πιστοποιητικά. Όχι. Έχουμε πει σε επιχειρήσεις, πάρτε τώρα πιστοποιητικά και τώρα ξαφνικά τους λέμε θα πληρώσετε. Αν έχετε αν θέλετε να ε, έχετε μεγαλύτερες εκπομπές. Η φιλοσοφία μας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας δεν έχει λειτουργήσει. Στα τελευταία 10 χρόνια, στα τελευταία 20 χρόνια έχει αυξηθεί η, η βιομηχανική πολιτική κατά 14,2 στη Γερμανία και η κατανάλωση ενέργειας έχει μειωθεί κατά 3%. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you for the comments. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Σημειώνουμε τα όσα ακούσαμε. Δεν ξέρω αν περιμένετε σχόλια από μας. Well, short and to the point, I'll say that. Ναι, ήσασταν ε, όντως ε, πολύ συγκεκριμένοι. Κύριε Βλάσακ, τι έχετε να απαντήσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλετε να απαντήσετε, δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε εδώ μαζί. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σημείωσα τα όσα άκουσα, αλλά θέλω να απαντήσω και σε κάποια σχόλια. Σίγουρα δεν αμφισβητώ το θέμα των ε, εκπομπών. Είναι στόχοι που έχουμε θέσει εμείς εξάλλου. Αλλά θα ήθελα να επιτρέψουμε περισσότερη ευελιξία για τις λύσεις που θα επιλέξουν ε, τελικά οι διάφορες χώρες. Δεν πρέπει δηλαδή να περιορίσουμε πολύ συγκεκριμένα. Δεν πρέπει να πούμε αεροδυναμική για παράδειγμα, γιατί ίσως υπάρχουν και άλλες λύσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης. Το ίδιο και για τα κίνητρα όσον αφορά την ανάπτυξη και την ε, καινοτομία. Σίγουρα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Όλα αυτά έχουν σχέση βέβαια και με την χρήση των κονδυλίων από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, συνεπώς, που πρέπει να εξεταστούν η ανάκτηση που λέτε ε, ενέργειας από τα ευρυδικά οχήματα. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν εδώ τα πράγματα και το βάρος και άλλα. Ευχαριστώ πολύ πάντως και προσβλέπω σε συνέχιση του διαλόγου και αν έχετε και σχόλια που θέλετε να μου στείλετε γραπτά, ευχαριστώ. 15 Ιουλίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 17 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ, στην Επιτροπή Ήτρε ψηφίζουν στις 14 Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τον Νοέμβριο. 15 Ιουλίου λοιπόν, 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στην επόμενη γνωμοδότηση που είναι της κυρίας Γκρίσμπεκ πρόταση κανονισμού για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Επιτροπή Μεταφορών με όρισε εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων στο πλαίσιο τη επιχειρησιακή συνεργασία που συντονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση τη επιχειρησιακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως λέει και ο τίτλος του κανονισμού, ήθελε, θέλησα να τον επαναλάβω, πρόκειται για ένα κείμενο που αφορά στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και που αφορά στην Επιτροπή Ελευθεριών επί της και εδώ με πολύ καλή θέση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διάσταση των μεταφορών είναι σχετικά περιορισμένη, μόνο η διάσταση ε, των μεταφορών αφορά μόνο την ε, αναζήτηση και την διάσωση αλλά και τον συντονισμό. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θέλησα να επικεντρωθώ γύρω από αυτές τις δύο πτυχές την ε, κατάρτιση των συνεργοφυλάκων για την προστασία των ατόμων βρίσκονται σε επικίνδυνο και ανταλλαγή προφοριών. Πρωτίστως σε ό,τι αφορά την αναζήτηση στη θάλασσα Προτείνω αυτές τις ρήτρες προστασίες όπως αυτές ε, καθορίζονται διάφορα πρωτόκολλα που ήδη ισχύουν για το παράνομο εμπόριο ε, των μεταναστών που είναι προσθήκη στην σύμβαση του ΟΗΕ για την ε, διεθνή εγκληματικότητα και την ε, μεταχείριση των ε, ατόμων που βρίσκονται στο σκάφος και την προστασία του σκάφους, του πλοίου, αλλά και του εμπορεύματος αυτού. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν την βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στην θάλασσα θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε και την ε, νομική κατάρτιση που προβλέπεται για την ανθρωπιστική βοήθεια και τις ε, ιατρικές πρώτες βοήθειες. Εξάλλου τα εμπλεκόμενα πλοία σε όλη φορά αυτήν την ε, ε, επιχείρηση θα πρέπει να έχουν όλα διάφορα kit ανθρωπιστικά και το οποίο περιέχουν και ιατρικά. Εγώ έχει τύχει να ανέβω σε σκάφος της Frontex που κάποια έχουν αυτά τα kit και κάποια όχι. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι τυποποιημένα αυτά τα kit και οργανωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στην θάλασσα και να προσπαθήσουν επίσης να έχουν και ιατρικό προσωπικό ε, στο πλοίο, επί του πλοίου. Αυτά χοντρικά για την κατάρτιση. Όπως είπα και αρχικά, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να οργανωθούμε αποτελεσματικότερα ή και να αυξήσουμε την ε, οργάνωση, την οργάνωση ανταλλαγής προφοριών ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τα εμπλεκόμενα μέρη όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της ε, ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Αυτή λοιπόν είναι μια ιδέα της διαλειτουργικότητας των συστημάτων εποτήρησης για να υπάρξει μια ε, παρακολούθηση που είναι απαραίτητη για την ε, θαλάσσια ναυσιπλοεία, για την προστασία των συνόρων και όλες τις δραστηριότητες ελέγχου ε, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Με αυτόν τον τρόπο οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι εποπτικές αρχές ε, θα μπορέσουν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα μειώνοντας ε, τις δαπάνες. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν βοήθειας και κατάρτισης, συλλογή των πληροφοριών για να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης και αναζήτησης. Ο οργανισμός θα πρέπει να φροντίζει να υπάρξει ένα κοινό, ένα κοινό πλαίσιο για την επιτήρηση του θαλασσίου τομέα της Ένωσης ε, και προτείνω λοιπόν στην έκθεση ο ρόλος του οργανισμού σε αυτό το ζήτημα να προσδιοριστεί στον κανονισμό συμπληρώνοντας τις διατάξεις που προέρχονται στην πληρώση που αφορά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης ε, Συνόρων Ευρωσύρου και καταλήγω λέγοντας Είδατε γιατί ο Πάπας ε, μετέβη στην ε, Λαμπεντούζα χθες προχθές και τόνισε την δυστυχία των ε, προσώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, πνίγονται και μετέβη επί για να δει πως έχει κατάσταση. Θα ήθελα να καταλήξω λοιπόν αναφερόμενοι σε αυτό το που υπόθηκαν γύρω αυτή την επίσκεψη του Πάπα και τρία χρόνια η νήσος Λαμπεντούζα ε, δέχεται χιλιάδες ε, μετανάστες, είναι ένας, μία, ε, ένα από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Θα υπερθυμίσω τον υποχρέωση για όλα τα σκάφη να βοηθούν όποια άτομα κινδυνεύουν στη θάλασσα και δυστυχώς μερικές φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της οδηγίας που αφορά στην είσοδο και παραμονή στο έδαφος της Ένωσης ε, παρανόμων και υπάρχει δυνατότητα να ε, κατηγορηθούν και να διωχθούν εάν ε, βοηθήσουν και προσφέρουν αρρωγή σε άτομα ε, μετανάστες που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί αυτό το κείμενο προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις καταστάσεις και το ε, θέμα της διάσωσης στην θάλασσα. Αυτά ε, συνάδελφοι, ελπίζω πως οι σκέψεις σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, οι κριτικές σας γιατί όχι θα περιοριστούν στην διάσταση της μεταφοράς της έκθεσης διαφορετικά. Θα πρέπει το ζήτημα να εξεταστεί περαιτέρω στην αρμόδια επιτροπή της Επιτροπής, δηλαδή την Επιτροπή Λίμπε. περίμενε το σχολιάζω, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ μέρους του ΕΛΚ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Γκρίσμπεκ για την συντήρηση που δεν είναι διόλου απλή, ακριβώς λόγω της δυσκολίας που ε, δημιουργεί η διάσταση ε, μεταφορών σε αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι οι προτάσεις της συναδέλφου πάνε προς την κατεύθυνση και παραμένουν ε, σταθεροί κάποιοι πυλώνες που έχουμε εμείς ως αρμοδιότητα της ΛΥΜΠΕ. Αν και, δεν, αν και δεν πρέπει να είμαστε τόσο άκαμπτοι, αλλά φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενίσχυση της δράσης της Frontex. Τα, τα πρόσφατα γεγονότα το, το καταδεικνύουν. Το βάρος της διαχείρισης αυτών των αφήξεων θα πρέπει να είναι αντικείμενο μια της συλλεγγύη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ενίσχυσης των κοινών εργαλείων και η Frontex είναι ένα από αυτά. Εγώ ε, δουλεύω πάνω σε κάποιες προτάσεις ε, ε, τροποποίησης και ολοκλήρωσης που αφορούν στις θαλάσσιες μεταφορές και που αφορούν την, τον ορισμό των γειτονικών περιοχών. Στη Μεσόγειο βασικά συχνά υπάρχει μια επικάλυψη ανάμεσα στις, στα ύδατα τα χωρικά μιας χώρας και τις λεγόμενες ε, γειτονικές χώρες που είναι ακριβώς δίπλα τις οικονομικές αποκλειστικές ζώνες ε, που αφορούν μια πιο εκτεταμένη περιοχή και μετά μιλάμε για τα εθνικά ύδατα στην την ανοιχτή θάλασσα. Λοιπόν, αυτές οι διαφορές, ε, μας αυτές οι διαφορές μάλλον προστίθεται και μια περαιτέρω κατανομή του θαλασσίου χώρου που αφορά τις ζώνες SAR, Search and Rest, που αφορά τις ιδιότητες ε, στις Frontex. Λοιπόν, ένας προκειορισμός και ορισμός αυτών των περιοχών και των σχετικών ευθυνών είναι απαραίτητο να γίνει, ειδικά αν ε, δούμε τη Μεσόγειο, όπου συχνά αυτές οι ζώνες, αυτή η υποδιέρεση, αυτή η κατανομή είναι ιδιαίτερα συγκεχημένη και οι ζώνες ε, επικαλύπτονται. Κατά τα υπόλοιπα, όπως είπα και πριν, το έργο της συναδέλφου είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε φυσικά στο πλαίσιο των αρμοδιών της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κύριε, ο το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο Γκρίσμπεκ για την ε, καλή της γνωμοδότηση. Η αντιμετώπιση της ε, διαθαλάσσης λαθρομετανάστευσης στην Μεσόγειο ιδιαίτερα μετά την ενίσχυση των χερσαίων συνόρων Ελλάδας και Τουρκίας, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως για τα πληρώματα των κρατών μελών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις που δυστυχώς όλο και πυκνώνουν εξαιτίας και όλης της εξέλιξης του κλίματος αστάθειας και ανάφλεξης στην, ε, στην ε, Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή δυστυχώς. Ε, ο στόχος της απόφασης του 2010 ε, όπως και τις πρώτες του κανονισμού που έχουμε μπροστά μας, είναι να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίε που έχουν εκφραστεί από κράτη-μέλη, από ακαδημαϊκούς, σχετικά με την τήρηση κάποιων θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα βέβαια στην ανοιχτή θάλασσα. Ε, είναι σαφές ότι τα πληρώματα και τα σκάφη που συμμετέχουν σε αποστολές αυτές οφείλουν να επιχειρούν με σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο για τα δικαιώματα ακόμα και όταν βρίσκονται σε ιδιαίτερα αντίξουες συνθήκες και απρόβλεπτες βεβαίως. Ε, συγκεκριμένα όμως όσον αφορά τα θέματα που άπτονται τουλάχιστον εμέσως της πολιτικής θαλασσίων μεταφορών πρέπει κατά τη γνώμη μας να διατηρηθεί η κατάλληλη ισορροπία αφενός μεταξύ της πληρότητας του κανονισμού και αφετέρου του ορθού διαχωρισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διεθνούς δικαίου. Τα ζητήματα της έρευνας και διάσωσης, καθώς και της αποβίβασης, καθορίζονται με επάρκεια εδώ και αρκετές δεκαετίες από τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις. Επομένως, θα πρέπει να εξετάσουμε στενότερα αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρμογή ή αλλίωσή τους, η οποία θα ήταν θεμητή μόνο για την καλύτερη επίτευξη του πρωταρχικού του σκοπού, την ασφαλή δηλαδή διάσωση και την αποβίβαση, και σε κάθε περίπτωση εντός του πλαισίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ο θεματοφύλακας εφαρμογής του εν λόγω Διεθνού Συμβατικού Πλαισίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Τέιλο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ πρώτης όψεως, αυτή η έκθεση δεν έχει μεγάλη εμβέλεια στον τομέα των μεταφορών, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Αλλά είμαστε σε μια κατάσταση πραγματικά σοκαριστική, όπου χιλιάδες άτομα πνίγονται στις προσπάθειές τους να φτάσουν τις ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πλοία τα οποία ψάχνουν για αυτούς τους επιζώντες και μετά γυρίζουν ε, πίσω ή φεύγουν παρά το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα σε κίνδυνο. Χαιρετίζουμε λοιπόν το άρθρο 9 το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό αντιμετωπίζοντας τα θέματα της έρευνας και τονίζοντας το στοιχείο της διάσωσης. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Συμφωνώ στο μεγαλύτερο μέρος με το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Γκρίσμπακ και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Πώς αυτή η πρόταση συνάδει και συμβαίνει συμβαδίζει με την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ε, πολιτική αυτή και τη χρηματοδότησή της. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας ε, δώσει εδώ μια απάντηση. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Επιτροπής εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκρίσπεκ για το σχέδιο γνωμοδότησής της και να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο για την ταχεία επεξεργασία του θέματος αυτού. Ίσως θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσω <clears throat> αναφερόμενος σε ένα θέμα που έθεσε ο κύριος Δανέλης σε σχέση με την συμβατότητα αυτών των ενεργειών με το Διεθνές Δίκαιο. Στις προτάσεις μας προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει συμβατό με το Διεθνές Δίκαιο, ιδίω για τις πράξεις έρευνας και διάσωσης μαζί με την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την έρευνα και τη διάσωση και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η πρόταση αυτή βασίζεται σε μια προσεκτική εξισορ... εξισορρόπηση συγγνώμη, μεταξύ του ελέγχου των συνόρων και των ενεργειών δράσεως και από την άλλη πλευρά των ε, στοιχείων συντονισμού, έρευνα και διάσωση που υπάρχουν ήδη στα κράτη-μέλη. Έχει διατυπωθεί η πρόταση με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό που έχουμε εδώ είναι η θέσπιση κριτηρίων για το τι πρέπει να ληφθεί υπόψη ως φάση εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή ο συναγερμό και οι πρώτες αντιμετωπίσεις όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος και στη συνέχεια οι επόμενες φάσεις συντονισμού θα περάσουν στο κέντρο έρευνας και διάσωσης της περιοχής όπου λαμβάνει η χώρα το επεισόδιο αυτό. Τώρα, η σύνδεση με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, όπως ε, ερώτησε ο κύριος Τέιλορ, το εργαλείο αυτό έχει σαν στόχο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη τα οποία λειτουργούν υπό το συντονισμό της Frontex αφεαυτού δεν είναι εργαλείο που έχει να κάνει με τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με το σχέδιο γνωμοδότησης, ιδίως για κάποια σημεία τα οποία έχουν αναφερθεί ήδη από την κυρία Γκρίσπεκ. Το πρώτο σημείο είναι η αναφορά στο κοινό περιβάλλον πληροφόρησης του Σέγγεν και η σχέση με τη Frontex. Θέλω να τονίσω ότι η Κομισιόν εργάζεται για την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας για το περιβάλλον του Σέγγεν που θα περιλαμβάνει και μια νομικού χαρακτήρα μελέτη και μια μελέτη των διαφόρων αρχιτεκτονικών μοντέλων ανταλλαγής πληροφοριών. Στο τωρινό στάδιο δεν έχει αποφασιστεί ακόμα σε σχέση με την διακυβέρνηση αυτού του περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, δηλαδή για το ποιος φορέας θα είναι αρμόδιος αν θα είναι η ΕΜΣΑ, η Frontex ή κάποιος άλλος φορέας. Ακριβώς γιατί υπάρχει το θέμα των νομικών αρμοδιοτήτων και της νομικής βάσης. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε κατατομής, μια κατατομής προσέγγιση και να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον ε, ανταλλαγής πληροφοριών μέσα από υπάρχοντα ίδια εργαλεία. Η δική μας εντύπωση όμως είναι ότι το τρέχον εργαλείο που αντιμετωπίζεται σε αυτή την πρόταση δεν θα πρέπει να προκαταλάβει τις συζητήσεις για το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών. Κάτι ακόμα που θέλω να αναφέρω είναι το θέμα της κατάρτισης για έκτακτη ιατρική βοήθεια και υποχρέωση να υπάρχουν ε, πρώτης, να υπάρχει εξοπλισμός πρώτης βοήθειας στα σκάφη. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο η νομική βάση που χρησιμοποιούμε σε αυτή την πρόταση μπορεί να καλύψει και τα θέματα της άμεσης ιατρικής βοήθειας και επομένως και την ιατρική κατάρτιση και θέματα όπως η παροχή εξοπλισμού για συγκεκριμένα σκάφη. Θα εξετάσουμε λοιπόν περαιτέρω το στοιχείο αυτό. Κάτι ακόμα το οποίο θα εξετάσουμε περαιτέρω εμπίπτει στην κατηγορία των ρητών προστασίας. Όταν υπάρχει μια πρόνοια αποζημιώσεως των σκαφών. Και αυτό θέλουμε να εξετάσουμε γιατί εδώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να αποδοθεί αποζημίωση δεν είναι σαφείς για μας και δεν είναι σαφές ποιος θα έδιδε αυτήν την αποζημίωση. Και επίσης η παραπομπή στο άρθρο 10 που δεν έχει να κάνει μονάχα με την αναχέτηση αλλά και την διάσωση φαίνεται ότι δεν θα ήταν καταρχήν ε, το κατάλληλο άρθρο. Αν έχετε περαιτέρω ερωτήματα είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκρισμπεκ. Έχετε να προσθέσετε κάτι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία απαντάει στις ερωτήσεις μου. Φυσικά θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε ξανά απόψεις. Να λάβουμε υπόψη μας την μελέτη αντικτύπου για παράδειγμα για την βελτίωση ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ποιος κάνει τι αλλά για την ε, ιατρική επίγουσα βοήθεια για αυτά τα ιατρικά kit ε, πάνω στα σκάφη και η κατάρτιση είναι κάτι σημαντικό. Θα έπρεπε να βρεθεί μια νομική βάση χωρίς δυσκολία. Τέλος πάντων, θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ βέβαια και τους συναδέρφους. Το θέμα των ορισμών των ζωνών είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω σε τι βαθμό έχει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει ανταποκριθεί νομίζω. Είμαστε εμείς η Επιτροπή Μεταφορών που πρέπει να δει το θέμα των ζωνών, τις διαφορές ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και οικονομικών περιοχών. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το θίξουμε, στη δικιά μας την έκθεση όχι. Εγώ θα έλεγα να συνεχίσουμε να το ψάχνουμε και αν ναι, τότε εννοείται είμαι στη διάθεσή σας για να δουλέψω και πάνω σε αυτό μια που είναι ακαθόδες πράγματι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας και με τις τροπολογίες θα επεξεργαστούμε παρετέρω το κείμενο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ναι, ευχαριστούμε. Κύριε Σίλη, έχετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, παρακαλώ, αλλά σύντομα. Ναι, ναι, ζητώ συγγνώμη κύριε Κρίσμπεκ. Δεν απάντησα στην ερώτησή σας για το θέμα των θαλασσίων ζωνών. Πράγματι. Σωστά. Δεν το θίγουμε το θέμα αυτό. Και ο λόγος είναι ότι είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας στα χώρια είναι θέμα χωρών ε, μελών δηλαδή και έχει να κάνει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Οι περιοχές διάσωσης όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Και αυτές καθορίζονται βάσει του Search and Rescue, της σύμβαση αυτής δηλαδή για την ε, διάσωση. Υπάρχει επικάλυψη μερικές φορές, με την πρόταση αυτή πάντως προσπαθούμε να σεβαστούμε τις θαλάσσιες περιοχές έτσι όπως καθορίζονται από τα κράτη-μέλη και να δουλέψουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε για δεύτερη φορά το λόγο. Πρόεδρος, καλώς. Υπενθυμίζω, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 11η Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Ψηφίζουμε στις 17 Σεπτεμβρίου και η Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη θα ψηφίσει τον Οκτώβριο. Συνεπώς, η πρώτη προθεσμία για τροπολογίες είναι η 11η Ιουλίου Παρασκευή. Πέμπτη, διορθώνει ο πρόεδρος, 12 το μεσημέρι, 11 Ιουλίου. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πολύ κρατάει, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι ευθυγράμμιση διαδρόμων Συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγηση τη πρόσκληση υποβολή προτάσεων για το 2012-2013. Ο κύριο Πακέτ. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο πολιετέ και το ετήσιο. Τέλο πάντων, έχετε το λόγο για να μα τα εξηγήσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να τα εξετάσουμε και τα δύο μαζί. Ναι, ναι, Αλλιώ θα χάσω την υπομονή μου. Ναι, ναι, κάντε το, ναι. Καλώ τότε, βεβαίω. Η ευθυγράμμιση διαδρόμων πρώτα, επιτρέψτε μου. Εδώ πέρα πρόκειται για ένα εγχείρημα που γίνεται από τους εισηγητές των ΤΕΝΤΗ και του ΣΕΦ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να διευκρινίσω λίγο την ευθυγράμμιση αυτή για την ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη με τα TNT. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν από το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και στη βάση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσει ότι η διάδρομη αυτή του ΤΕΝΤΗ και οι άλλοι εννέα για την, ε, το συνδέοντα στην Ευρώπη δεν συγκλίνουν πάντα δεν ευθυγραμμίζονται πάντα και γι' αυτό προσπαθούμε να τους ευθυγραμμίσουμε γεωγραφικά. Το πλεονέκτημα της άσκησης αυτής ευθυγράμμισης είναι βέβαια πολιτικό, γιατί έχουμε έτσι μία ομάδα διαδρόμων που καλύπτει τις πολυτροπικές μεταφορές και δίνεται έτσι και μεγαλύτερη προβολή Συγχρόνως όμως προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε και την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη ε, αξία, γιατί έτσι οι εμπορικοί διάδρομοι υποφελούνται από όλες τις πολιτικές και από την διαχείριση ημέν των δε. Είναι κάτι που προωθείται και εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά διαπιστώνουμε και τα κρατημέλη δηλαδή ότι είναι κάτι πολύ ε, θετικό. Χωρίς λοιπόν να μπω στις λεπτομέρειες της ευθυγράμμισης αυτής, νομίζω και η Νέσα Γιάλα και ο κύριος Δικέ θα σας μιλήσει για τα πορίσματα των τριμερών διαλόγων, αλλά αν δείτε το παράτημα για την διευκόλυνση της στην Ευρώπη, θα δείτε ότι οι διάδρομοι που περιγράφονται στο παράρτημα έχουν μειωθεί από 10 στους 9 γιατί έχει υπάρξει κάποια συγχώνευση και γράμμιση έκανε αλλαγέ επίσης. Οπότε στο παράρτημα επίσης αυτό θα βρείτε και την περιγραφή, την νέα ...και την περιγραφή των εμπορικών μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων. Όταν αρχίσουν να ισχύουν τα TNT, δηλαδή και η διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη στα τέλη τη χρονιά, θα έχετε περισσότερα στοιχεία και οι εμπορικοί αυτοί ε, διάδρομοι θα διευκρινιστούν περισσότερο. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που όσον αφορά και τα TNT και του σιδηροδρόμους, η διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη πρέπει να επιβεβαιωθεί. Και αύριο ελπίζουμε στην Κορεπέρ να γίνει αυτό. Άπαξ και έχει γίνει θα έχουμε κάνει και ένα μεγάλο βήμα στην πολιτική μας για τις εμπορικές μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων. Τώρα δύο λόγια για τα τεντή και για την φετινή διαδικασία επιλογής. Έχουμε όντως ε, μία μπροσούρα για το ετήσιο πρόγραμμα και άλλη μία για το πολιετές. Γιατί γίνεται μια ετήσια δουλειά για τα κατά προγράμματα και μια πολιετής μπροσούρα για τα υπόλοιπα προγράμματα. Την τελευταία φορά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κάποια χρηματοδότηση που παραμένει. Και γι' αυτό μάλλον μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα επανέλθουμε εδώ με ένα επιπλέον πρόγραμμα εργασίας. Αλλά το αφήσουμε αυτό για μετά το καλοκαίρι. Προς το παρόν είναι η τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 1,5 δις ευρώ συνολικά και για το ετήσιο και για το πολιτές. Άρα είναι υψηλή η χρηματοδότηση, η οποία θα οδηγήσει σε πέντε φορές παραπάνω συνολικό ποσό επενδύσεων. Και τα δύο, και το τίσιο και το πολιτές, και θα τα δείτε αυτά στα φυλαδιά μας, υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ και μερικές μέρες, θα δείτε όλα τα δεδομένα για, την, για τις μεταφορές ανά μέσο θα δείτε ότι υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις στα TNT σε σχέση με τα τελευταία 6 χρόνια. Και θα δείτε ότι υπάρχουν σημαντικές προτεραιότητες που στηρίζουν τις μεταφορές είτε για την ΕΤΜΕΣ είτε για την διαχείριση ενέργειας κυκλοφορίας και βέβαια για τους, ε, τις διαδρομές της θαλάσσιας τρεις-τέσσερις τορυδικές προτεραιότητες σε προγράμματα είναι για την πρόθεση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Οι υποδομές και η χρηματοδότηση, δηλαδή των καθαρών μεταφορών, περιλαμβάνονται εδώ. Υπάρχει επίσης και το στοιχείο στο ετήσιο πρόγραμμα της συνεργασίας ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Προσπαθούμε να υπάρξει ένα μείγμα ε, κονδυλίων από τα κράτη-μέλη και από επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Ελπίζουμε έτσι να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και τους μελλοντικού διαδρόμους. Υποδομές, συνεπώς, αλλά πάντα ανάλογα με τις προτεραιότητες μας και τις πολιτικές μας. Τώρα για το πολιτες πρόγραμμα. Το κύριο που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι η επιλογή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε πέντε φορές παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα που χρειάζονται χρηματοδότηση. Δυστυχώς όμως οι επενδύσεις είναι περιορισμένες από τα κράτη-μέλη. Σημαίνει βέβαια αυτό συγχρόνως ότι η επιλογή γίνεται δύσκολη. Και μερικές φορές αναγκαζόμαστε να περιορίσουμε τα προγράμματα ανάλογα με την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στην Ευρώπη και ανάλογα με το αν πιστεύουμε ότι πράγματι μπορούν να αποδώσουν γρήγορα μια που είναι η τελευταία χρονιά των προγραμμάτων. Αυτά είναι τα δύο κριτήρια λοιπόν τα οποία ακολουθήσαμε για να κάνουμε την επιλογή αυτή από προτάσεις που όπως σας είπα ήταν πέντε φορές παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Για 1,5 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το πρώτο σημείο. Έχω μονάχα δύο ή τρεις ερωτήσεις ή σχόλια. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Κομισιόν γιατί μας έχει δώσει ήδη τα στοιχεία σχετικά. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι άμεσες επιπτώσεις στις εμπλεκόμενες χώρες και κατά πόσο αυτή η από κοινού θέση ε, βοήθησε τις συγκεκριμένες αυτές χώρες, ιδίως τις χώρες αυτές που έχουν προβλήματα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις χρονικές στιγμές, αν για τα διάφορα κράτη-μέλη έχει προταθεί ένα χρονοδιάγραμμα για να μπορέσει να γίνει η ενσωμάτωσή τους προοδευτικά και επί ποιας βάσης έχει δημιουργηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και τρίτον Υπάρχει μια διαδικασία η οποία έχει προταθεί για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα συγχρησιμοποιηθεί η ίδια για τους διαδρόμους ή προβλέπεται μια διαφορετική διαδικασία. Και δεύτερον, το δεύτερο ερώτημα, δεν είχα αρκετό καιρό να αναδειφίσω το έγγραφο αυτό, γιατί σήμερα μοναχαρία διανεμήθηκε. Θα το διαβάσω στις καλοκαιρινές μου διακοπές, όμως σας το υπόσχομαι. Έχω ένα ακόμα ένα απλό ερώτημα για τις ε, πολιετής προσκλήσεις βλέπω την, ε, τον, ένα, ένα, τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας μεταξύ αυτών. Μα είμαστε σε μια κατάσταση που είναι φανερό ότι οι ενιαίοι ευρωπαϊκοί εθέρες δεν έχουν εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη, ή δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν για πολιτικούς λόγους, πώς συνδέεται αυτό με τις επενδύσεις που αναφέρατε με την τωρινή πρόταση της Κομισιόν, την νέα της πρόταση για τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες. Οι επενδύσεις οι οποίες θα θεωρηθούν σύμμορφες είναι σύμμορφες και με το δεύτερο δεύτερη εκδοχή της πρότασης Κομισιόν ή μόνο με την πρώτη πρόταση Κομισιόν ή δεν υπάρχει καμία απολύτως σύγκρουση μεταξύ των δύο προτάσεων της Κομισιόν. Μπορείτε να μου δώσετε και γραπτά στοιχεία αν θέλετε. Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις πληροφορίες που μας έδωσε και επίσης τις πληροφορίες που μας έδωσε για το, τα σχέδια που υπευλήθηκαν για το τελικό στάδιο της χρονικής περίοδου 2007-2013. Είπατε ότι μετά το καλοκαίρι θα υπάρξει ένα πρόγραμμα, δεν κατάλαβα ακριβώς τι θα κάνει αυτό το πρόγραμμα. Θα υπάρχει χρηματοδότηση ή όχι για αυτό το νέο πρόγραμμα. Δεύτερον, μπορεί να μας πει ίσως η Κομισιόν αν είχε περισσότερο, περισσότερη χρηματοδότηση, πόσα προγράμματα παραπάνω θα μπορούσε να έχει εγκρίνει. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να εντοπίσουμε καλύτερα το κατά πόσο υπήρχαν προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν πέραν αυτών τα οποία δεν είχαν καμία προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν τελικά υπήρχαν προγράμματα ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας που δεν μπόρεσαν να, χρηματοδοτηθούν. Θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ να ξέρουμε πόσα προγράμματα μπορούσαμε στην πράξη να χρηματοδοτήσουμε, γιατί αυτό θα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε σχέση με τον πολιετή προϋπολογισμό, τι δημοσιονομικής προοπτικές δηλαδή. Και τέλος, σε αυτή τη διαδικασία ε, υποβολής προσφορών σχεδίων, δεχόμαστε προγράμματα σε αιτήσιο επίπεδο και πολιετή που έχουν να κάνουν με την ε, μεταρρύθμιση των πολιτικών αυτών πώς θα λειτουργήσει η Κομισιόν, πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα προγράμματα που είναι στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ της παλιάς και της νέας προγραμματικής περίοδου. Και τέλος έχουμε κάποια εθνικά σχέδια τα οποία παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή που είναι σε κατάφορη σύγκρουση και αντίφαση με την διευκόλυνση Connecting Europe. Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει η Κομισιόν αυτά τα εθνικά σχέδια τα οποία έχουν χαρακτήρα αντίθετο με αυτό του Connecting Europe. Ο κ. Κόλτσεκ. Έχω να πω τα Κύριε Πακέ, αντιληφθήκατε ότι η Κεντρική Ευρώπη λείπει από αυτά τα προγράμματα. Ενώ σε φορά το νότο της Ευρώπης υπάρχουν δεκάδες ε, προγράμματα που έγιναν δεκτά. Φαίνεται πως ε, οι κυβερνήσεις ε, των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης δεν τους ζητήθηκε καν να συμμετάσχουν. Είναι που βάλουν προτάσεις τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα της, των αεροπορικών συντέσεων. Βλέπω ότι για την κεντρική Ευρώπη τα πράγματα δεν λειτουργήσαν, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, οι κυβερνήσεις δεν ενεργούν όπως θα έπρεπε. Εάν θέλουμε λοιπόν να βελτιωθούν τα πράγματα στην κεντρική Ευρώπη, π.χ. οι Αυστριακοί δεν έλαβαν τις απαραίτητες αποφάσεις και ε, να πω κάτι για τον ε, ενιαίο ε, ευρωπαϊκό εθέρα και για τα προγράμματα απλούστευσης φαίνεται ότι τα πράγματα στην Κεντρική Ευρώπη δεν είναι έτοιμα να εξελιχθούν. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ. Ε, Ευχαριστώ. <clears throat> ναι, κοίταξα τώρα το έγγραφο αυτό για την ετήσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Στη σελίδα τώρα 79 έχω ένα πρόβλημα. Είναι μια μελέτη. Μια νέα γραμμή μεταξύ Καβάλας και τα χωτάει. και εδώ φαίνεται ότι αυτό έχει κλείσει και η Ελλάδα χρηματοδοτεί ήδη αυτή τη γραμμή. Τι θα γίνει τώρα αν κλείσει αυτή η γραμμή γιατί συνεχίζει και πηγαίνει στο Σβίλεγκρατ και στην Τουρκία στη συνέχεια θα κατασκευαστεί αυτή, είναι σε επίπεδο μελετών τι ακριβώς θα συμβεί με αυτή τη γραμμή. Και το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ έχουμε πει πάντα για τη γραμμή Λιών Τωρίνο που που δεν θα κοστίσει 2, 12 εκατομμύρια αλλά 26 δισεκατομμύρια συγγνώμη και υπάρχει μια μελέτη στη Γαλλία που είπε ότι πρέπει να κλείσουμε αυτή, αυτό το εγχείρημα δεν έχει κανένα νόημα έχουμε ήδη πολλά τρένα υψηλής ταχύτητας σίγουρα μέχρι το 2030 δεν θα έχει τελειώσει αυτή η γραμμή είναι κάτι που θα σταματήσει, λέμε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αλλού, δεν μας ενδιαφέρει και άλλες μελέτες έχουν προτεραιότητα γιατί αυτό δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί με το 2030 παρά το γεγονός ότι υπήρχε απόφαση των κρατών μελών. Καλό είναι να θέλουμε να τα κάνουμε όλα, αλλά τα σχέδια τελικά χρηματοδοτικά δεν έχουν ευοδοθεί. Τι θα κάνετε, θα καταλήξουμε λοιπόν με, σε ένα σωρό μελετών οι οποίες δεν θα πραγματοποιηθούν τελείως. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τις μελέτες εκεί που υπάρχει πράγματι μια δυνατότητα να υλοποιηθούν όλα αυτά και να μπορέσει να υπάρξει μια κατασκευή για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Όχι μόνο άσκηση επιχάρτου, όχι στο χώρο των ονείρων. Θέλουμε όλα αυτά τα σχέδια να γίνουν πραγματικότητα. Αλλιώ δεν έχει νόημα να τα κάνουμε. Ο κύριος Έρτου. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και για τον φορέα των διευρωπαϊκών δικτύων που αναλαμβάνει αυτό το έργο και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα σχέδια τα οποία έχουν επιλεγεί. Από τα 134 έχουμε 89 ε, τα οποία επελέγησαν. Αυτό το οποίο εγώ βρίσκω ιδιαίτερα θετικό είναι ότι δίνουμε τη σωστή έμφαση γιατί ο, το κέντρο βάρους είναι τα σιδηροδομικά σχέδια και τα σχέδια εσωτερικών υδατίνων οδών και η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφοράς. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτά να είναι στο κέντρο των προσπαθειών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και αυτό είναι ο σωστός δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι αν δούμε τα πράγματα για το μέλλον, εδώ θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η πίεση αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ για τις χώρες συνοχής που είναι προσδιορισμένα για αυτές τις χώρες και επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την, ε, τα εγχείρηματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο φιλόδοξοι στα θέματα αυτά και θα ήταν χρήσιμο και παρακαλώ την Κομισιόν να σκεφτεί καλύτερα για το θέμα αυτό γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αιτιολόγηση και η αξιολόγηση για την επιλογή αυτών των, των σχεδίων ίσως θα μπορούσε κανείς να εξευγενήσει ακόμα περισσότερο την επιχειρηματολογία για τους λόγους για τους οποίους επιλέγονται ακριβώς αυτά τα σχέδια. Σίγουρα θα υπάρξει και μεγαλύτερη πίεση όταν είναι όλο και περισσότερα τα προγράμματα τα οποία υποβάλλονται θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για την Κομισιόν και θα είναι ευφυέ και λογικό αν η Κομισιόν δίνει μια καλύτερη επιχειρηματολογία για τους λόγους που επιλέγει ορισμένα προγράμματα και σχέδια. Έχω επίσης και ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς την Κομισιόν για το 31066 αν δεν έχω καταλάβει αν έχω καταλάβει καλά πρόκειται για 7 δισεκατομμύρια ευρώ που θα πάνε στην εταιρεία Nissan Motor 7,3 εκατομμύρια συγγνώμη, για να χρηματοδοτήσει τους σταθμούς αυτούς επαναφόρτισης στα πλαίσια του σχεδίου 13 που είναι η σύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Ιρλανδίας. Το, το ερώτημα μου είναι κατά πόσο εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης 50% και αν αυτό είναι απαραίτητο για την ε, βιομηχανία δημιουργία σταθμών επαναφόρτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως προβλέπετε εδώ. Και το δεύτερο μου ερώτημα είναι... αν αυτή η σταθμή επαναφόρτησης της ε, Nissan ε, είναι πολλαπλών, ε, πολλαπλών προτύπων, δηλαδή δέχονται διάφορες μορφές πριζών για τα... έχουν διάφορες μορφές ε, για πρίζες αυτοκινήτων και επίσης αν στις προσπάθειες, στις προσπάθειες στη... για πρόθεση των εναλλακτικών εταιριών η Κομισιόν θέλει να προωθήσει μονάχα ένα τύπο για πρίζες, για φορτιζόμενα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κατά το οποίο μου φαίνεται να μην συνάδει με τις προτάσεις της Κομισιόν εν γέννη. Και επίσης για το σχέδιο Swiftly Green εδώ δεν έχω καταλάβει περί πρόκειται και θα ήθελα να μας εξηγήσετε καλύτερα σε τι συνίσταται αυτό το Swiss Green το σχέδιο και για ποιο ακριβώς λόγο θα δοθεί η χρηματοδότηση. Αυτά θέλω να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ έχω πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία έχω. Φυσικά πρέπει να δούμε προσεκτικά το τι είναι το κάθε ένα από αυτά τα σχέδια. Ο κύριος Κράμερα αναφέρθηκε σε ορισμένα σχέδια. Εγώ έρχομαι από την ε, Βόρεια Ευρώπη και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τα ναυτικά θέματα, ιδιαίτερα όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον ναυτικό χώρο και σχέδια όπου υπάρχει χρηματοδότηση, τους νέους ε, καθαριστές για, τα, για τις εκπομπές διοξιδίου του θείου ή για το energy bunkering, την ε, αποθήκευση ενέργειας και για τη σύνδεση με την Τάλιν. Πιστεύω ότι εδώ η βασική αρχή είναι ότι όλα αυτά τα σχέδια τα οποία έχουν προτεραιότητα είναι αυτά τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει τις γρηματοδόσεις και μπορεί κανείς να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσει η υλοποίησή τους. Αυτό είναι που θελήσαμε εμείς, θέλουμε να γίνουν ε, ενέργειες οι οποίες μπορούν να καρποφορήσουν. Σωστό είναι αυτό, θα ήταν πολύ καλό να είναι έτσι. Ευχαριστώ. Oh, okay. Dominic. Dominic. Dominic. Ναι. Σύντομα, γιατί μιλάμε και για αιτήσια προγράμματα, μιλάμε και για ευθυγράμμιση διαδρόμων. Τώρα βέβαια με... Στα συγγνώμη από την κυρία Λασέντερ Σέντερ, τους άλλους ε, εισηγητές, αλλά θέλω να ξέρω, οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εισηγητές πρέπει να μου πούνε, κανένα πρόγραμμα τελικά από αυτά που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν πρέπει να εξαφανιστεί. Και δεύτερον, η ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα να παραμείνουν, να μην αλλάξουν τα κριτήρια δηλαδή. Δεν λέω ότι απαντάει αυτό στην ερώτηση του Ματιέ. Φαντάζομαι ότι θα απαντήσει σε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι εδώ δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το οποίο έχει ήδη δουλέψει και ψηφίσει η Επιτροπή μας και για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πρόεδρος, καλώς. Μια από τις δυσκολίες εδώ είναι ότι έρχεστε, μα τα αφήνετε αυτά και μετά φεύγετε. Αλλά βλέπετε άμα δώσετε ένα χάρτη σε έναν πολιτικό, τι κάνει, αμέσως κοιτάζει τα δικά του. Λοιπόν, ίσω για το μέλλον θα έπρεπε την διευκόλυνση συνδέοντα για την Ευρώπη, για παράδειγμα, και τα ευρωπαϊκά δίκτυα να τα έχουμε εκ των προτέρων, ώστε να τα έχουμε διαβάσει και όταν έρχεστε εδώ να μπορούμε να σας ρωτήσουμε. Γιατί ωραία. Και την προηγούμενη φορά ήρθατε, μας κάνατε την παρουσίασή σας, μας δώσατε τα βιβλιαράκια σας, μετά τα διάβασα και είπα αύριο να πάρει, αν τα είχα διαβάσει πιο πριν και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τα διάφορα προγράμματα, και εδώ θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις σας, σύντομα, αλλά ό,τι επιπλέον πληροφορίες θέλετε, Ευχαριστώ. είμαστε στη διάθεσή σας στη συνέχεια. Αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, το οποίο είτε επιλέχτηκε είτε δεν επιλέχτηκε, ευχαρίστως να συζητήσουμε μαζί σας γι' αυτό. Ό,τι πληροφορίες θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Με τη σειρά θα πάρω τις ερωτήσεις. Ντομινίκ Ρίκε, ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε για τους διάφορους διαδρόμους εμπορικής μεταφοράς και διευκόλυνσης. Ναι, οι επιπτώσεις είναι σημαντικές της ευθυγράμμισης, θέλω να πω. Έχουμε επιπλέον διαδρόμους ή επιπλέον τμήματα σε ήδη υπάρχοντες εμπορικούς διαδρόμους σιδηροδρόμων. Και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, καλύπτονται όλες οι χώρες μέλη συστηματικά και για όλους τους νέους εμπορικούς διαδρόμους τώρα υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από το 2016 μέχρι το 2020 ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο φόρτος είναι διαχειρίσιμος κυρίως για τις χώρες εκείνες μέλη που θα έχουν επιπλέον εμπορικούς διαδρόμους Συνοδρομικούς πάντα. Σίγουρα στο τελευταίο στάδιο του εγχειρήματο για την ευθυγράμμιση ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά φροντίσαμε να μην υπάρχουν εξαιρέσει και να καλύπτονται όλε οι χώρε μέλη και υπάρχουν στοιχεία για όλου του διαδρόμου. Βέβαια, υπάρχει χωριστή νομοθεσία, γιατί εδώ δεν περιλαμβάνεται το περιεχόμενο, αλλάζουν τα παραρτήματα, δημιουργούνται νέοι διάδρομοι, αλλά ο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται η διάδρομη αυτή είναι κάτι διαφορετικό. Για τους ε, ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες. Ετοιμάστηκε το πρόγραμμα πριν έχουμε το δεύτερο πακέτο υπήρχαν ήδη οι προτάσεις. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει κάτι που δείχνει έλλειψη συνοχής. Ευχαριστώ όμως οι συνάδελφοι από τη Διεύθυνση για τις Αεροπορικές Μεταφορές να σας ενημερώσουν παρετέρω. Νομίζω ότι όλοι υποφελούνται και από τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Όσον αφορά την ε, κεντρική Ευρώπη, πάντως θα επανέλθω σε εσάς αν συμφωνείτε, θα ρωτήσω τους συναδέρφους και θα σας ενημερώσω παρετέρω. Τα ποσά που δεν καλύπτονται. Πρόκειται για το πολιετές πρόγραμμα. 1,3 δισεκατομμύρια είναι διαθέσιμα. 5,7 δις θα έπρεπε να είχαμε για να καλύψουμε όλα τα προγράμματα. Και κρατήσαμε μόνο τα πιο όριμα προγράμματα, αυτά επιλέξαμε. 4,3 δις θα χρειαζόμασταν για όλα αυτά. Για τα καλά δηλαδή, 4,3 δισεκατομμύρια θα χρειαζόμασταν. Και έχουμε 1,3. Παρετούμαστε δηλαδή από 3 δισεκατομμύρια συγχρηματοδότηση χρηματοδότηση, επειδή δεν υπήρχε επαρκή χρηματοδότηση. Βέβαια, στο ετήσιο τα ποσά είναι πολύ πιο χαμηλά. Είμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο με το ποσό που τελικά είμαστε σε θέση να διαθέσουμε. ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν επιπλέον ε, κονδύλια διαθέσιμα σύντομα όταν ένα πρόγραμμα έχει καθυστερήσει, όπως το έχουμε ήδη συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή σας, και δεν μπορούν έγκαιρα να προχωρήσουν οι δραστηριότητες, δεν δίνεται η χρηματοδότηση από τη δικιά μας την πλευρά, μπορεί συνεπώς να επανέλθει στο πρόγραμμα και άρα να γίνει μια μικρή πρόσκληση υποβολής ε, προτάσεων μετά το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να επιλέξουμε επιπλέον προγράμματα. Πράγματι υπάρχουν ε, σε μερικές χώρες λίγα προγράμματα. Αυτό το βλέπουμε και από τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και γιατί, γιατί τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι πολύ χαμηλά προκειμένου η δίκηση να επιλέξει τα διευρωπαϊκά δίκτυα αντί για τα κονδύλια συνοχής. Και γι' αυτό, μετά από πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, έφτιαξε αυτό το παράθυρο για τα δέκαδη. Άρα υπάρχει συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και να στηριχθούν έτσι τα διευρωπαϊκά δίκτυα και στις 28 πια χώρες μέλη. Όσον αφορά μελέτες, Έχουμε λιγότερες μελέτες. Βέβαια προσοχή γιατί οι μελέτες μπορεί να είναι και πιλωτικά προγράμματα. Οπότε μπερδευόμαστε στην ορολογία μέσα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Οπότε το 20-25% των ε, μελετών δεν είναι απαραίτητα σε χαρτί, μπορεί να είναι πιλωτικά προγράμματα. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν πρέπει να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι εφόσον χρηματοδοτούνται οι μελέτες, χρηματοδοτούνται στα πλαίσια μιας αξιόπιστης προοπτικής για το μέλλον. Θα επανέλθω πάντως για αυτό το ελληνικό πρόγραμμα, ε, Μάκη, να σου απαντήσω παρετέρω. Όπως και σε προηγούμενα προγράμματα, έτσι και τώρα θέλουμε βιώσιμες ε, μεταφορές, τρόπους μεταφοράς και αυτό είναι κάτι που κυριαρχεί και στα ετήσια προγράμματα και στα πολιετή. Είναι κριτήριο επιλογής δηλαδή. Γι' αυτό χρησιμοποιούν και τα κράτη-μέλη τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και θα τελειώσω με το πρόγραμμα καινοτομία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, πολλές βρίζες. Απλώς θέλουμε να δείξουμε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο, οπότε η χρηματοδότηση ακόμα και για την βιομηχανία του 50% δικαιολογείται. Πάντα όμως παίρνουμε και μαθήματα από το παρελθόν. Για το Swiftly Green είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για το μέλλον μαζί με τις κατευθυντήριες γραμμές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο έχει υπογραμμίσει τις βιώσιμες και πράσινες μεταφορές για τους διαδρόμους αυτούς. Οπότε πρόκειται για μια απόδειξη του πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω με αυτούς τους ε, corner corridors. Από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή σας ό,τι παρατέρω πληροφορίες θέλετε, αν θέλετε για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο, ευχαρίστω να σας ενημερώσουμε παρετέρω. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, θα περάσουμε τώρα στη συνεδρία των θυρών. Όσοι λοιπόν δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται, ας αποχωρήσουν.